θεωρώ ότι είναι κατεπίγουσα ανάγκη να κινηθούμε προς την κατεύθυνση μιας πρώιμης ε, δεύτερης ανάγνωσης. Βοηθήστε μας λοιπόν για να καταλήξουμε από κοινού σε μια καλή διαπραγματευτική θέση. Αν δεν το καταφέρουμε αυτό και περάσουμε στην κανονική διαδικασία της δεύτερης ανάγνωσης, η επιρροή του Κοινοβουλίου θα είναι σαφώς μικρότερη. Και δεν μπορούμε να υποθέσουμε ότι το Συμβούλιο αυτόματα θα υιοθετήσει τις ε, θέσεις του Κοινοβουλίου. Τη δική τους θέση θα έχουμε επιτάπητος και θα συζητήσουμε. Και θα μπορούμε να θέσουμε, να υποβάλουμε τροπολογίες, αλλά θα πρέπει να τις περάσουμε με ειδική πλειοψηφία. Και κοιτώντας πώς έχει η κατάσταση και τα συμφέροντά μας, θα πρέπει να σας πω ότι μάλλον χαμένοι θα βγούμε παρά κερδισμένοι. Γι' αυτό λοιπόν σας παρακαλώ, σας θερμοπαρακαλώ να βοηθήσετε κι εσείς προκειμένου να περάσει αυτό το θέμα έτσι και όσο πιο πολλά θέματα διευκρινίσουμε με το Συμβούλιο, όσο πιο πολλά θέματα ε, λύσουμε, τόσο πιο εύκολη θα είναι η συνέχεια. Και είμαι πεπισμένη ότι πέρα από τα όρια των ομάδων θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Γι' αυτό λοιπόν απευθύνω αυτή την έκκληση και πέρα από τα όρια των ομάδων. Να πετύχουμε μία συμφωνία με το Συμβούλιο, η οποία θα αποβεί προς όφελος και των ζώων αλλά και της υγείας των ανθρώπων. Βρισκόμαστε εν το μέσο των εργασιών μας να διευκρινίσω ποιε θα είναι οι επόμενε μεγάλε συναντήσει μα. Ο επόμενο τριμερή διάλογο την 5η 12 Νοεμβρίου. Και πάντα συμμετέχουν, πάντα είναι προσκεκλημένοι οι σκιώδει και αν δεν μπορέσουν να παρευρεθούν, ε, μπορώ να λάβω γραπτό τις θέσεις που θέλουν να εκπροσωπήσω. Ίσως στις 20 Νοεμβρίου να λάβουμε κοινή θέση του Συμβουλίου και ο επόμενος τρομερής διάλογος ενδεχομένως 24-25 ε, Νοεμβρίου, 1η Δεκεμβρίου και το Συμβούλιο Γεωργίου, Γεωργίας. Αν ε, μας δώσετε και την έγκρισή σας και εσείς ε, Πρόεδρε, 14 και 15 Δεκεμβρίου. Έχουμε πολλά να κάνουμε λοιπόν μπροστά μας. Υπάρχουν και θέσεις στις οποίες το Συμβούλιο δεν ε, συμφωνεί καθόλου. Έχει λάβει το Συμβούλιο, δηλαδή, τη δική μας θέση, αλλά δεν έχω λάβει οποιαδήποτε αντίδραση, άρα δεν ξέρουμε κατά πόσο συμφωνεί ή όχι. Είμαι αισιόδοξη πάντως και θεωρώ ότι στο σημείο αυτό πρέπει να ευχαριστήσω και τους εκπροσώπους της ειδική Προεδρίας. Από τον Ιούλιο ήταν πολύ χρονοβόρα και πολύ εντατική αλλά και πάρα πολύ καλή η συνεργασία μας τελικά. Ευχαριστώ πραγματικά θερμά όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ κυρία Γέγγελ. Νομίζω ότι έχουν προχωρήσει πολλοί εργασίες και είμαι πεπισμένος ότι αυτή η έκκληση που κάνετε θα γίνει δεχτή από όλους τους βουλευτές. Ξεκινάμε τώρα τη συζήτηση. Μα ζητάνε διάφοροι το λόγο. κυρία Σάρμπο είναι η πρώτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξανά ευχαριστήσω και εγώ την ε, κυρία Γέγκλη για την πολύ καλή συνεργασία. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τους άλλους συναδέλφους και εισηγητές Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση των διαπραγματεύσεων έχουμε προχωρήσει. Καταφέραμε να, προχωρήσαμε, για... να προχωρήσουμε γιατί συζητήσαμε και συμφωνήσαμε. Είναι σημαντικό να έχουμε μια κοινή θέση στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να πετύχουμε σχεδόν όλα όσα επιθυμούμε σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες γιατί η κυρία Γέγκελ μας παρουσίασε λεπτομερώς τα πράγματα. Το μόνο που θέλω να σας πω είναι ότι φτάσαμε σε συμβιβασμό ε, για διάφορα άρθρα, παραδείγματος χάρη τον τρόπο σφαγής των ζώων για να μειώσουμε τα, τα προβλήματά τους, τα βασανά τους και τα είδη υπό Άλλο άρθρο. Αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα σοβαρά σημεία τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε στις επόμενες ε, συναντήσεις μας για να φτάσουμε σε μια κοινή θέση, σε μια συνεννόηση. Επαναλαμβάνω ότι στηρίζουμε πλήρως αυτή την ιδέα της ευημερίας των ζώων και ελπίζω πραγματικά να φτάσουμε σε καλά αποτελέσματα. Ευχαριστώ ακόμα όλους ε, όσους συμμετείχαν ε, δεύτερη φορά και νομίζω ότι θα, θα ξανασυζητήσουμε αυτά τα θέματα. Δεν έχει τελειώσει η συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Μαγκίνε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να, ευχαριστήσω την κυρία Γέγκλε για τον τρόπο που χειρίστηκε το δοσχέ αυτό, γιατί έθεσε με πολύ αποτελεσματικό τρόπο και πολύ ειλικρινή και άμεσο τα επιχειρήματα αυτά για την ευημερία των ζώων. Πρόσφατα έλαβα πολλά mail από την επιστημονική κοινότητα που εκφράζει ανησυχίες για την οδηγία. Δεν ξέρω αν ε, οι επιστήμονες είναι ενημερωμένοι για τις τελευταίες εξελίξεις που μας περιέγραψε η Ελίζαμπεθ. Ανησυχούν για τα άρθρα 8 και 16 της πρότασης οδηγίας. Και ίσως ε, στη δευτερολογία της η Ελίζαμπεθ θα μπορούσε να κάνει την ε, διάκριση μεταξύ βασικής και εφαρμοσμένης τεχνολογίας και τον περιορισμό με βάση τους στόχους της έρευνας και με βάση το θέμα της ευημερίας των ζώων. Γιατί η επιστημονική κοινότητα πραγματικά ανησυχεί με το θέμα αυτό. Ενδιαφέρεται για την ευημερία των ζώων, αλλά θα πρέπει να βρεθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ των αναγκών της επιστημονικής κοινότητας και των αναγκών της ευρύτερη κοινωνίας, αλλά και τα... την ευημερία των ζώων. Και ελπίζω αυτό να το προσέξει εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Ελίζα, την οποία ευχαριστώ θερμά για την προσφορά της. Κυρία Πόλσεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ την κυρία Γέγκλε, η οποία έκανε μια θαυμάσια δουλειά. Καθόλου εύκολη δεν ήταν το έργο της, γιατί υπήρχαν πάρα πολλές διαφωνίες και πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ των ε, έτσι, φανατικών ακτιβιστών και κάποιων επιστημόνων. Παραμένουν βέβαια ως κρεμή κάποια θέματα, τα οποία ανέφερε η κυρία Γέγκλη. Παραδείγματος χάρη ο έλεγχος. Από τότε που εξελέγει στο Κοινοβούλιο, ξέρω ότι γράφονται οι νομοθεσίες, περνάνε οι νομοθεσίες, ψηφίζονται νόμοι, αλλά μετά δεν γίνεται τίποτα. Ο έλεγχος λοιπόν είναι κεντρικό στοιχείο. Εν συνεχεία, η συζήτηση για τα μεγάλα πρωτεύοντα, τους, πίθη, τους πίθηκους, τους μεγάλους πίθηκους. Εκεί το Συμβούλιο έχει παρουσιάσει μία σαφή απέτηση όπου λέγεται ότι όλες οι ασθένειες όλες οι αρρώσεις θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο να μπορούν να αποτελούν αντικείμενο έρευνα. Παραδείγματο χάρη ο διαβήτη. Εγώ νομίζω ότι το Συμβούλιο δεν έχει αυτό το δικαίωμα. Υπήθηκε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ε, σε έρευνα όταν πρόκειται για νευρολογικές ασθένειες. Όταν μιλάμε για έρευνα ε, στον εγκέφαλο, για τους νευρολογικούς διαβιβαστές. Εκεί η χρήση των πυθίκων μπορεί να είναι αναγκαία, αλλά όχι στον τομέα ασθενειών που είναι αρκετά συνηθισμένες, ε, γνωστές και όπου υπάρχουν άλλες λύσεις. Νομίζω ότι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι στο φαρμακευτικό τομέα είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιούνται αυτά τα ζώα. Παραδείγματο χάρη, ε, γυναίκες όπως εγώ που έχουν πατήσει τα 70 και που καταπίνουμε τις χούφτες στα φάρμακα για να αποφύγουν το διαβήτη, ναι, θα πρέπει να έχουν σωστές λύσεις, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να γίνεται ε, εις βάρος της υγείας των ζώων. Um, Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Γέγκλε για τον τρόπο που χειρίστηκε τις διαπραγματεύσεις και κυρίως ε, για τη στενή συνεργασία που είχε σε πρόωρο στάδιο της διαπραγμάτευσης με τους σκιώδεις ηγητές. Περιμένουμε χρόνια ολόκληρα αυτή την ε, νομοθεσία και θέλουμε να είναι αυστηρότερη από την ισχύουσα νομοθεσία για να μπορέσει και η επιστημονική κοινότητα να βρει εναλλακτικού τρόπους και να μην χρησιμοποιεί μόνο ζώα στην έρευνα. Σε ό,τι φορά τη χρήση των πρωτευόντων θηλαστικών, θα πρέπει να είναι πολύ περιορισμένη και ε, έχουμε φτάσει λεπτομέρειες διαπραγμάτευσης για θέματα ιδιαίτερα προσφυλή, όπως είναι ο τρόπος αδειοδότησης ε, για τις ε, δοκιμές. Στο άρθρο 2, για παράδειγμα, πιστεύουμε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν αυστηρότερους κανόνες για όλες τις πτυχές αυτής της νομοθεσίας δεν θα πρέπει τα κρατημέρια να υποχρεώνονται να υποβαθμίζουν τις προδιαγραφές τους εξαιτίας αυτής της ε, κοινοτική νομοθεσία. Θα πρέπει να υπερισχύουν οι εθνικές αυστηρότερε ε, διατάξεις. Επίσης θέλουμε η αναθεώρηση να γίνεται κάθε μία διετία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά τη χρήση των ε, πρωτευόντων θηλαστικών που δεν είναι άνθρωποι και επίσης να βρεθούν κάποιοι μέθοδοι αντικατάστασης εναλλακτική χρήση. Δεν θέλουμε ε, χαμηλές προδιαγραφές ή αόριστη διατύπωση, γιατί είναι θέμα κοινού και δημόσιο ενδιαφέροντος. Όλοι ε, γνωρίζουν τι τεράστια είναι τα λόμπι για τα θέματα αυτά και θα πρέπει να δείξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι ανησυχεί για τα θέματα αυτά και θέλει ακρίβεια και αυστηρότητα. Δεν θα πρέπει να είμαστε χαλαροί και δοτικοί. Συμφωνώ και με την πρόταση της κυρίας Γέγκλε για την αύξηση του αριθμού των ελέγχων. Νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε συμφωνία με το Συμβούλιο για να εξασφαλίσουμε τουλάχιστον δύο ελέγχους το χρόνο. Για το άρθρο 37 πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει μία και του διοντολογικού στοιχείου. Να γίνει μία διοντολογική ηθική αξιολόγηση του προγράμματος και όχι μόνο μια αξιολόγηση του προγράμματος χωρίς το επίθετο δεντολογικό ή ηθικός. Δεν μπορούμε να επισέλθουμε σε όλες τις λεπτομέρειες τώρα. Ελπίζω να συνεχιστεί η ηθικο δεν μπορουμε να επισελθουμε σε ολες τις λεπτομερειες τωρα ελπιζω να συνεχιστει η πρόοδο στι συζητήσει με το Συμβούλιο. Στόχος μας φυσικά είναι η επίτευξη συμφωνίας, αλλά όχι εις βάρος ε, των θέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όχι υποχωρώντας. Θέλουμε αυστηρή κοινοτική νομοθεσία για το θέμα αυτό, ώστε οι επιστήμονες να χρησιμοποιούν ε, εναλλακτικού τρόπους πειραματισμού και να μην καταφεύγουν στη χρήση πειραματοζώων συστηματικά. Ο Λουίς Άλβες. Καπόλα Σάντος, συγγνώμη. Όλοι γνωρίζουμε πόσο ευαίσθητο είναι αυτό το θέμα, πόσο λεπτό και πόσο φορτισμένο συγκινησιακά, γιατί όλοι αγαπούμε τα ζώα. Μερικοί έχουμε <laughs> ζώα που είναι μέλη της οικογένειάς μας σχεδόν. Και γι' αυτό ε, ασχοληθήκαμε με το θέμα αυτό διεξοδικά στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία. Είχαμε πολύ ωραίες ακροάσεις, προσπαθήσαμε να ακούσουμε όλα όλο το φάσμα των απόψεων. Είχαμε διαβουλεύσει και με πολλούς επιστήμονες και πιστεύω ότι η θέση στην οποία καταλήξαμε είναι πολύ ισορροπημένη. Και ευελπιστώ ότι το νέο κοινοβούλιο με τους νέους βουλευτές που δεν συμμετείχαν στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις θα είναι ακόμη πιο φιλόδοξο και θα τελειοποιήσει τις σημαντικές συμβαστικές προτάσεις που διαμορφώσαμε τους προηγούμενους μήνες. Η κυρία Γέγκλε είναι πεπειραμένη ευρωβουλευτής, με ιδιαίτερες ευαισθησίες και με πλούσια γνώση για το θέμα αυτό και πιστεύω ότι θα πρωτοστατήσει τις διαπραγματεύσεις και θα τις ε, χειριστεί με επιδέξιο τρόπο. Το ίδιο και οι υπόλοιποι συνάδελφοι που συμμετέχουν στη διαπραγματευτική ομάδα. Είναι πολύ δύσκολο το έργο, το αντιλαμβάνομαι, γιατί όλοι υφιστάμεθα τεράστιες πιέσεις, αρκεί κανείς ε, να ανοίξει τα mail του, του ταχυδρομείου του ηλεκτρονικού για να διαπιστώσει πόσες πιέσεις και πόσα mail λαμβάνει για το θέμα, αυτά, για το θέμα αυτό και ελπίζω μετά με την ε, υιοθέτηση αυτής της έκθεσης να καταλήξουμε σε ευρεία συνενετική θέση. Ευχαριστώ και ευχαριστώ πως έκανε και σκιώδη συγκεκριά μας την κυρία Γέγκλε για την προσφορά της. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ελίζα Μπατκέγκλα εξ ονόματος της ομάδας μου και εξ ονόματος όλων των συνεργατών μου να σας ευχαριστήσω για την καλή συνεργασία και για την καλή έκθεση στην οποία καταλήγουμε. Θα ήθελα να θέσω κάποια θέματα. Αν δεν βρούμε μία εύλογη ρύθμιση, δεν ε, προστατεύουμε ουσιαστικά τα ζώα, γιατί ξέρουμε ότι μπορεί να μετακατασταθεί και η επιστήμη και η έρευνα και αυτό δεν είναι προς το συμφέρον των εν λόγω ζώων, όταν τα πειράματα δηλαδή αυτά ε, μεταγκατασταθούν εκτός Ευρώπης. Δηλαδή, αν δεν είναι εύλογη η ρύθμιση που θα επικρατήσει, θα έχουμε προβλήματα γι' αυτό λοιπόν αυτό το καυτό θέμα δεν ενδείκνεται για κομματικές διαφορές και διαφωνίες. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να διαμορφωθεί μια διαφορετική κατάσταση προκειμένου να μην βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου ως κοινοβούλιο δεν θα μπορούμε να επηρεάσουμε την ε, θέση που θα επικρατήσει. Γι' αυτό λοιπόν εγώ και η ομάδα μου υποστηρίζουμε τη θέση της Ελίζα Μπεθ Γέγκλε. Ξέρει και γνωρίζει τέλεια το θέμα και θα πρέπει λοιπόν να την υποστηρίξουμε προς το συμφέρον των ζώων. Ευχαριστώ, Άλμπερτ. Κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και εγώ την κυρία Γέγκλε για την εξαιρετική αυτή έκθεση. Στην Αυστρία το 2005 πέρασε ένας πάρα πολύ σύγχρονος ε, νόμος για την προστασία των ζώων με πολύ αυστηρά μέτρα σε σχέση με το διεθνές προσκήνιο. Και γι' αυτό θεωρώ ότι η πρόταση για τους ε, αυστηρούς ελέγχους είναι πραγματικά πάρα πολύ σωστή. Γι' αυτό λοιπόν απευθύνω έκκληση για την διαμόρφωση μεγάλη πλειοψηφία υπέρ τη έκθεση αυτή στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ και τελευταίο ομιλητή, ο κύριο Γιάρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την κυρία Γέκλη για την πολύ καλή έκθεση και εγώ επίσης θα χαιρόμουν αν ε, θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε πέρα από τα όρια των ομάδων για το θέμα αυτό. Γιατί αυτό αποτελεί και τη σωστή αντιμετώπιση, αν θέλετε, για το πρόβλημα. Θα ήθελα, μετά από αυτά που είπε και ο κύριος Ντές, να προσθέσω δύο στοιχεία Συμμετείχα σε σχετικές κοινοβουλευτικές ε, επιτροπές του Γερμανικού Κοινοβουλίου και πάντα με ανησυχούσε το εξή: ότι καταρχάς ο νομοθέτης ο ίδιος, εμείς δηλαδή, θα πρέπει να προσέξουμε ως νομοθέτες να μην ε, δημιουργούμε νέα ενάψματα για πειραματόζωα. Να αναφέρω για παράδειγμα το πρόγραμμα REACH, το οποίο έχει έναν εύλογο πυρήνα, αλλά να κοιτάξουμε τα στατιστικά στοιχεία στη Γερμανία αυξήθηκαν ε, οι δοκιμές σε πειραματόζωα. Και εγώ πρέπει να σας πω ότι με ανησυχεί ο αριθμός των ε, δοκιμών που προέρχονται από το πρόγραμμα REACH. Άρα, ως νομοθέτης πρέπει να προσέξουμε, να μην δημιουργήσουμε νέες ε, αφορμές για δοκιμές. Και το δεύτερο, όπου έχω μεγάλες επιφυλάξεις, είναι οι διάφορες έρευνες που θα καταστήσουν ε, περιτές τις δοκιμές στα ζώα για παράδειγμα, σε αιμοριακό ή κυταρικό επίπεδο. Νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει αρκετά σε επίπεδο, στο επίπεδο αυτό στην Ευρώπη και εδώ παρουσιάζεται το πρόβλημα το εξή. Οι χώρες προσπαθούν να αναγνωριστούν αυτές οι δοκιμές. Και συνάδελφε Γέγκλε, εκεί θα ήθελα να αναφέρουμε στην έκθεση ότι απευθύνουμε έκκληση προς ε, τα κράτη-μέλη για να ενθαρρυνθούν να προχωρήσουν με τα κυταρικά αυτά, με τις κυταρικές αυτές και ε, μοριακές δοκιμές, οι οποίες ενδεχομένως να καταστήσουν ε, περιττές τις δοκιμές σε περιγραμματόζωα. Καλώς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους έλαβαν μέρος στη συζήτηση και να συγχαρώ και εγώ θερμά την κυρία Γιάγκλα και καλή σας επιτυχία στις περαιτέρω διαπραγματεύσεις με βάση το χρονοδιάγραμμα που μας προδιαγράψατε. Θέλετε να δευτερολογήσετε για να ολοκληρώσουμε αυτό το σημείο της της διάταξης, Ελίζαπεθ. Ναι, ευχαρίστω, Πρόεδρε. Να επαναλάβω ότι ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους. Κάποιες παρατηρήσεις τις οποίες δικαίως θίξατε είναι, για παράδειγμα, στοιχεία επί των οποίων δεν έχει συμφωνήσει ακόμα το Συμβούλιο σε ό,τι αφορά τις έρευνες, τους μετέπειτα ελέγχους, κυρία Πάουλτσεν. Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι θα υπερφορτωθεί με τους ελέγχους αυτούς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει ελέγχους από τα εθνικά συστήματα και κάνει η ίδια μόνο σπραδικούς ελέγχους. Αυτό είναι το σύστημα που επικρατεί. Θα πρέπει να το συζητήσουμε ενδεχομένως. Θεωρώ λοιπόν ότι οι ευνηδιαστικοί αιτήσιοι έλεγχοι μπορούν να αποτελέσουν το σωστό μέσο και θα πρέπει να συζητήσουμε επίσης και τα θέματα που αφορούν τα μεγάλα πρωτεύοντα και θα πρέπει να βρούμε συμβιβασμό ο οποίος ενδεχομένως να πονέσει και κάποιους όπου και πάλι θα πρέπει να ξεκινήσουμε με βάση την έκθεση, ε, την έκθεση του Κοινοβουλίου. Ε, το ίδιο και για τις διαδικασίες έγκρισης αντιοδότησης. Αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε, το επαναλαμβάνω, είναι να μην ε, επανέλθουμε στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό το καταδεικνύουν άλλωστε και κάποιες από τις παρατηρήσεις σας. Ε, να πω επίσης στους συναδέλφους ότι οι τροπολογίες οι οποίες αφορούν, ε, μάλλον που αφορούν πληροφορίες που μας δίνουν οι ενώσεις προστασίας των ζώων, θεωρώ ότι ισχύουν αλλά βρισκόμαστε σε φάση διαπραγματεύσεων και δική μου βάση είναι το κείμενο το οποίο έχουμε εγκρίνει, το οποίο έχουμε ψηφίσει και να σας διαβεβαιώσω ότι συζητώ με όλες τις ενώσεις προστασίας των ζώων που θέλουν να μου μιλήσουν, ακόμα και αν είναι πολύ χρονοβόρα αυτή η διαδικασία. Γνωρίζω λοιπόν τι γίνεται σε αυτό το επίπεδο και ρώτησα όλες τις ενώσεις τις τελευταίες εβδομάδες τι ακριβώς επιθυμούν. Και με μία μοναδική εξαίρεση ενός ατόμου μίας ένωσης μόνο, μόνο ένα άτομο ήθελε δεύτερη ανάγνωση λοιπόν. Όλοι οι υπόλοιποι, όλες οι υπόλοιπες ενώσεις ήταν ικανοποιημένες με το εύρος της απόφασης και με τον την οδό που θέλω να ακολουθήσω, κοιτώντας την οδηγία του 86, την παλιά οδηγία. Να το συνειδητοποιήσουμε αυτό, ότι ούτε εμείς, ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούμε να προωθήσουμε μία καινούργια οδηγία. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Κοιτάξτε, είναι το πρώτο βήμα που κάνουμε μετά το 1986. Δεν πρέπει να το δυσκολέψουμε παραπάνω από ότι χρειάζεται. Και έχουμε τα τρία R που αναφέρονται στο κείμενο. Μείωση, αντικατάσταση και αυτό απέχει παρασάγκας και βελτίωση. Απέχουμε λοιπόν παρασάγκας από αυτά που φανταζόμαστε στην αρχή. Η Γερμανία, η Αυστρία, έχουν ε, περάσει νόμους για την προστασία των ζώων πολύ αυστηρούς. Η Γερμανία το έχει κατοχυρώσει και στο Σύνταγμα μάλιστα. Λοιπόν, τα κράτη-μέλη αυτά δεν μπορούν να επαναχωρήσουν σε σχέση με τους νόμους τους. Θα πρέπει να δούμε ποιος διασφαλίζει την καλύτερη προστασία των ζώων, και παράλληλα προοδεύει περισσότερο από κάθε άλλον σε θέματα έρευνας. Είναι πολύ σημαντικά τα θέματα αυτά. Σας ευχαριστώ και πάλι και σας παρακαλώ να με υποστηρίξετε για να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία. E- σας ευχαριστώ. Χαίρι στις μέρη της υποστήριξης ε, και εμπιστοσύνης της Επιτροπής μας. Χαρητήρια ήταν πολύ σημαντική προσφορά σου και ελπίζω να διεκπεριωθεί αυτό το θέμα, αν όλα πάνε καλά, πριν τα Χριστούγεννα. Περνούμε στο σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης τώρα. Την αξιολόγηση και εκτίμηση του σχεδίου δράσης για την καλή μεταχείριση των ζώων κατά την περίοδο 2006-2010. Το σχέδιο δράσης για την ευημερία των ζώων θα ολοκληρωθεί. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε ένα νέο σχέδιο δράσης, μια και θα εκπνεύσει το προηγούμενο και φυσικά θα πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση κατάσταση προκειμένου να χαραχθούν οι κατευθυντήριε γραμμέ για το μέλλον. Γι' αυτό και η Επιτροπή μα αποφάσισε να καταρτήσει έκθεση πρωτοβουλία για το θέμα αυτό. Η συγγήτριά μα είναι η κυρία Μάριτ Πόλσεν, στην οποία θα δώσω και το λόγο προκειμένου να μα διαφωτίσει. Έχει το λόγο Μάριτ. Tack, herr ordförande och ärade σας ευχαριστώ. Θα συνεχίσουμε ουσιαστικά την προηγούμενη συζήτηση που είχαμε με την κυρία Γέγκλε, γιατί για τα ίδια ζώα μιλάμε και τα ίδια προβλήματα. Και το θέμα είναι εξίσου λεπτό και ευαίσθητο. Λίγα είναι τα θέματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που προκαλούν τόσο έντονες ε, και σφοδρές αντιδράσεις. Το θέμα της ευημερίας και της καλής μεταχείρισης των ζώων είναι ένα από τα θέματα αυτά. Άλλα θέματα είναι λιγότερο ευαίσθητα. Αυτό όμως είναι ιδιαίτερα λεπτό γιατί έχουμε να δώσουμε λόγο απέναντι στους πολίτες μας, στους, εκλε... στους ψηφοφόρους μας. Το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό και ο τρόπος με τον οποίο μια κοινωνία μεταχειρίζεται τα ζώα δείχνει πόσο πολιτισμένη και ανεπτυγμένη είναι. Δεν έχουμε βέβαια πολλές αρμοδιότητες για το θέμα αυτό. Και έχουμε φυσικά τα κατοικίδια ζώα όπως είναι οι γάτες, οι σκύλοι, οι παπαγάλοι. Αλλά πολλοί πολίτες θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δικαιούται να λάβει αποφάσεις για τα κατοικίδια, για παράδειγμα. Αλλά εδώ εμείς δεν ενδιαφερόμαστε για τα κατοικίδια, ενδιαφερόμαστε κυρίως για τα ζώα εκτροφής, τα ζώα της κτηνοτροφίας. Και θα πρέπει να επικεντρωθούμε και σε κάποια δευτερεύοντα θέματα. Δηλαδή στις οικονομικές πτυχές και σε κάποια γραφειοκρατικά ζητήματα που απορρέουν από την προστασία των ζώων. Για παράδειγμα, κάποιες προδιαγραφές που θα πρέπει να ισχύουν για τα σφαγεία. Αλλά ο γεωργός ή ε, ο κτηνοτρόφος είναι αυτοί που σε τελική ανάλυση έχουν το ηθικό βάρος, το οικονομικό βάρος και έχουν όλα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ε, σωστή μεταχείρισης των ζώων. Οπότε ο Γιώργος και ο κτηνοτρόφο βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της συζήτηση. Στην έκθεσή μου προσπάθησα να χωρίσω το θέμα σε τρεις κατηγορίες. Καταρχήν, κάνω μια ανάλυση του κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταπεξήλθε στις δεσμεύσεις και τις υποσχέσεις της. Επίσης λαμβάνω υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2006 που είχε εκπονήσει η κυρία Γέγκλε. Και κάνω μια αξιολόγηση της εφαρμογής αυτού του ψηφίσματος και το κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έλαβε υπόψη και αν ε, έλαβε υπόψη και την ε, δηλωμένη τότε βούληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προωθήσει αυτό το θέμα. Έγινε μια προσπάθεια να συμπεριληφθούν και κάποιες νέε πτυχές στο θέμα τη καλής μεταχείρισης των ζώων, με βάση το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλά παρά τα έντονα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, κόφευσε. Και φαίνεται ότι έχουμε απομακρυνθεί αρκετά από το ψήφισμα του 2006. Εμείς, παρόλο που είμαστε νέο κοινοβούλιο, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τη συνέχεια του κοινοβουλευτικού έργου και θα πρέπει να επιμείνουμε στις απαιτήσει του προηγούμενου ψηφίσματος. Ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προβλέπει ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι νέες τεχνολογίες και τα νέα επιστημονικά πορίσματα και ανακαλύψεις. Και υπάρχει και ένα σχέδιο που ασχολείται με την καλή μεταχείριση και την ευημερία των ζώων και δίνει κάποιους επιστημονικούς δείκτες για την ανάπτυξη των ζώων, για τη μεταχείριση των ζώων. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να γίνει εύκολα αντιληπτό το θέμα. Τα κοτόπουλα, για παράδειγμα. Γνωρίζετε ότι αγκιστρώνουμε τα κοτόπουλα σε μία μακριά αλυσίδα, σε τσιγκέλια, ε, πριν τα αναισθητοποιήσουμε. Και υπάρχει και μία κάμερα που ε, μαγνητοσκοπεί τα πόδια των ε, κοτόπουλων και κινητοποιείται ένα συναγερμό όταν διαπιστωθεί ότι τα, τα πόδια τους έχουν κάποιες πληγές. Βέβαια, όταν η εκτροφή έχει 10.000 κοτόπουλα, κάποιοι κοτόπουλα πέθαναν ε, από σύνθλιψη. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτός ο έλεγχος. Αλλά φροντίζουμε ώστε ο αριθμός των τραυμάτων να είναι περιορισμένος, να μην έχουμε πολλές πληγές. Αν βρεθούν πολλές πληγές στα πόδια των κοτόπουλων, ενεργοποιείται ο συναγερμός. εκτός από την ε, κλασική νομοθεσία προστασίας της ευημερίας των ζώων, δεν χρειαζόμαστε και τέτοιους επιστημονικούς δείκτες. Γιατί τέτοια μέτρα είναι πολύ πιο συγκεκριμένα και ακριβή και χρειαζόμαστε και αξιόπιστα στοιχεία για να κάνουμε αξιολόγηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάστηκε πολύ σκληρά τα τελευταία χρόνια και παρόλα αυτά δεν μας ικανοποίησε σε όλα μας τα αιτήματα, αλλά έχει μείνει χρόνος ακόμη και μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταλήξει στα επιθυμητά αποτελέσματα. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθεται και καρτερεί, γιατί αναμένεται η νέα συνθήκη και φυσικά θα σχηματιστεί και η νέα Επιτροπή. Γι' αυτό το μέλλον είναι κάπως αβέβαιο. Πάντως, με την Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ έχουμε πολύ στενή συνεργασία και πολύ καλή. Και εκεί δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, ούτε ε, κολλήματα στην ε, επίτευξη μιας συμφωνίας. Τι μπορούμε να πούμε λοιπόν για το μέλλον. όλοι οι σκιώδεις συζητητές θα πρέπει να συνεργαστούν μαζί μου ώστε να καθορίσουμε από κοινού τα βασικά στοιχεία της θέσης μας και τις ε, μελλοντικές μας απαιτήσεις ε, για το σχέδιο δράσης μετά το 2010. Βέβαια δεν είναι, δυνατόν, δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν όλες οι επιθυμίες και όλες οι απαιτήσει. Εμείς θα επικεντρωθούμε στα πιο ουσιαστικά ζητήματα της κοινοτική νομοθεσίας, της μελλοντικής κοινοτική νομοθεσίας για την σωστή μεταχείριση των ζώων. Το θέμα των ελέγχων, των ελέγχων εφαρμογής είναι πάρα πολύ σημαντικό. αλλά θα πρέπει να δει και κάποια συνέχεια. Έχει νόημα να συντάξουμε μια νέα οδηγία για τη μεταφορά των ζώων όταν γνωρίζουμε ότι ο έλεγχος αυτής της μεταφοράς είναι προβληματικός. Γιατί δεν εφαρμόζουν όλα τα κράτη με τον ίδιο τρόπο αυτόν τον έλεγχο και αυτές οι διαφορές υπάρχουν. Υπάρχουν και νέες προηγμένες τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Το σύστημα δορυφορικής πλοήγησης, για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ε, εποπτεία της μεταφοράς των ζώων, για τη διάρκεια της μεταφοράς, τη θερμοκρασία του οχήματος, ε, το ποσοστό υγρασίας, όλα αυτά τα στοιχεία μπορούν να καταγραφούν. Γιατί η πληροφορική σήμερα είναι σε θέση να επεξεργαστεί μια σωρία τέτοιων στοιχείων. πολλές φορές η εξονυχιστική ανάλυση της μεταφοράς ε, ισχυρίζονται μερικοί ότι υποβαίνει βάρος της ε, προστασία της ιδιωτικής σφαίρας των οδηγών. Δεν ευσταθεί όμως αυτό το επιχείρημα γιατί το GPS χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της μεταφοράς των φορτηγών για παράδειγμα. Εκεί γνωρίζουμε πότε κάνει στάση για να πάει στην τουαλέτα ο οδηγός της Νταλίκας. Δεν ισχυρίζεται κανένας όμως ότι αυτό ε, παραβιάζει την ιδιωτική του σφαίρα. Άλλωστε, ο οδηγός που πραγματοποιεί τη μεταφορά είναι σε όρο εργασίας. Δεν παραβιάζει την προσωπική του ζωή με το να, ελέγχεται, να ελέγχονται οι συνθήκες μεταφοράς μέσω του συστήματος δορυφορικής πλοήγησης είναι σαν να παρακολουθούμε με κάμερα του ταξιτζίδε. Δεν υποστηρίζει κανένα ότι παραβιάζει η ιδιωτική του ζωή. Υπάρχουν λοιπόν λύσει που μα δίνουν νέε τεχνολογίε που όμω δεν εφαρμόζονται. Επίση θα πρέπει να βρούμε ποια είναι τα κεντρικά στοιχεία, τα πιο ουσιαστικά ζητήματα. Θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε ορισμένες βασικές επιθυμίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να μην ξεχνάμε ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες που μας δίνουν οι νέες τεχνολογίες. Γιατί αυτός ο τομέας είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την Επιτροπή Γεωργίας. Πιστεύω ότι ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των ζώων έχει τη θέση του στο κέντρο της συζήτηση για τις αξίες της νέας κοινή γεωργικής πολιτικής. Το θέμα της ευημερίας και της καλής μεταχείρισης των ζώων αποτελεί το πιο στέρεο επιχείρημα για να διαφυλάξουμε τα πιο σημαντικά στοιχεία της κοινή γεωργικής πολιτικής. Μία κτηνοτροφία που θα μας δίνει υγιή ζώα. Θα αποτελεί ουσιαστικό κλάδο της δημόσιας υγείας της Ένωσης, γιατί ζώα που έχουν υποστεί κακή μεταχείριση, που χρειάζονται αντιβιωτικά και φάρμακα, επηρεάζουν αρνητικά τη δημόσια υγεία. Είναι μεγάλος ο αριθμός των φαρμάκων και των αντιβιωτικών που χρησιμοποιούνται στην κτηνοτροφία, κάτι που οδηγεί σε όλο και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στα μικρόβια. Δεν θα πρέπει να υπάρξει σύγκρουση μεταξύ του αιτήματο ευημερία των ζώων και του αιτήματο εξασφάλιση τη δημόσια υγεία. Θα πρέπει στο μέτρο του δυνατού να περιοριστεί η χρήση αντιβιωτικών και φαρμάκων στη γεωργία και την κτηνοτροφία. Α σκεφτούμε την υγεία των παιδιών μα, την υγεία των εγγονών μα. Γιατί να μην διοργανώσουμε ένα σεμινάριο για τις νέες επιστημονικές ανακαλύψεις και τα νέα ερευνητικά πορίσματα. Προτείνω να διοργανώσουμε ένα τέτοιο σεμινάριο τον Ιανουάριο-το Φεβρουάριο και από εκεί να τροφοδοτήσουμε τη συζήτησή μας. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό να διοργανώσουμε ένα τέτοιο σεμινάριο, αλλά το προτείνω και ελπίζω να γίνει. Όλο και νέε τεχνολογικές εξελίξεις υπάρχουν, γιατί να μην τι εκμεταλλευτούμε. Σας ευχαριστώ. Ε, Paulson, Ευχαριστώ την κυρία Πόλσον. Και τώρα θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Υπάρχουν διάφορε παρεμβάσει. Η κυρία Γιάνγκη. Καταλαβαίνετε βεβαίω ότι υπάρχει μια συνάφεια ανάμεσα στο προηγούμενο σημείο και σε αυτό εδώ. Επομένω, πρώτη και καλύτερη κυρία Γέγκλε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ πάρα πολύ και την κυρία Πόλσεν, την εισηγήτρια. Ναι, υπάρχει συνάφεια και σε αυτή την στρατηγική για την προστασία των ζώων 2006 έως 2010 είχαμε θέσει την απέτηση αυτή. Μετά την οδηγία για, την, για τα πειραματόζωα. Ανταποκρίθηκε λοιπόν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είχαμε συζητήσει τα θέματα αυτά. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κυρία Πάλουσεν για την ε, δουλειά σας, την οποία έχω μελετήσει. Θεωρώ ότι είναι και πολύ καλό και πολύ σημαντικό να στηριχτείτε σε αυτή την έκθεση, γιατί ήταν τότε πάρα πολύ αμφιλεγόμενη η έκθεση αυτή και μάλιστα μας κόστησε πάρα πολύ χρόνο, αλλά τελικά πετύχαμε ένα καλό αποτέλεσμα. Ένα σημείο θα ήθελα να επισημάνω και να επιστήσω προσοχή. Το σημείο το οποίο δικαίως και πολύ σωστά δείξατε κι εσείς η ίδια. Η έκθεση πρωτοβουλίας αυτής ε, αναφέρεται στα ζώα που χρησιμοποιούνται στη γεωργία. Έχει συζητηθεί και στην έκθεση για το 2005-2006 και τότε ως κοινοβούλιο καταλήξαμε μετά τη συζήτηση στο ότι εμείς ως κοινοβούλιο μπορούμε να θέσουμε τον όρο αυτό για, άλλα, για όλα τα ζώα. Να πούμε δηλαδή ότι εντάξει, ναι, συμφωνούμε, είναι καθήκον μας ε, να ρυθμίσουμε το θέμα των ζώων εκτροφής, αλλά όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη έκθεση, είναι ηθική μας ε, η υποχρέωση προς όλα τα ζώα. Δεν μπορούμε αυτό να το μεταβιβάσουμε προς την επιστήμη έχουμε ευθύνη για όλα τα ζώα. Το είχα πει αυτό και το θυμήθηκα γιατί μας είπατε ότι το θέμα των ζώων είναι σημαντικό και αμφιλεγόμενο. Αλλά γιατί δηλαδή ο σκύλος επειδή είναι ζώο συντροφιάς περνάει καλύτερα, θα τον βάζω σε ένα μικρό κλουβάκι και τον αφήνω 10 ώρες ε, στο αεροπλάνο. Δηλαδή δεν διαφωνώ, τα ζώα εκτροφής, ε, η απόδοση είναι το αντικείμενό μας, αλλά θα πρέπει νομίζω να συμπεριληφθούν όλα τα ζώα. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε τώρα με την κυρία Γκαρσία Περές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και την κυρία Πόλσεν για την έκθεσή της μπορώ να τη βεβαιώσω εκ των προτέρων για την αμέριστη συνεργασία της ομάδας μου για το θέμα αυτό. Χθε μιλούσαμε για την πολιτική της ποιότητας, σήμερα για την πολιτική της ευημερία. Όλα αυτά δείχνουν ότι θέλουμε ένα ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο που δεν θα περιορίζεται στην παραγωγή, αλλά θα σέβεται αυστηρές προδιαγραφές και διατάξεις για την παραγωγή αυτή. Κάτι που προϋποθέτει η προσπάθεια των γεωργών και των παραγωγών μας. Αλλά το αποτέλεσμα θα δίνει προστιθέμενη αξία στα γεωργικά προϊόντα. Επειδή μιλήσαμε για το μελλοντικό πρόγραμμα δράσης, σχέδιο δράσης, πιστεύω ότι πριν προβούμε στην εκπόνηση του μελλοντικού σχεδίου, θα πρέπει να αξιολογήσουμε το προηγούμενο και το κατά πόσο υλοποιήθηκαν οι στόχοι και έγιναν σεβαστοί πέντε πυλώνες του προηγούμενου σχεδίου δράσης για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να προσαρμοστούμε με βάση τις νέες προκλήσεις. Αναφέρθηκαν οι εφαρμοστέοι κανόνες σε θέματα καλής μεταχείρισης και ευημερία, αναφέρθηκαν τα θέματα έρευνας, η συμπερίληψη κάποιων δικτών ευημερία, μεγαλύτερη συμμετοχή. Θα πρέπει αυτούς τους πέντε πυλώνες ε, να τους ελέγξουμε, να δούμε εφαρμόστηκαν σωστά. Μήπως θα χρειαστεί συμπερίληψη νέων δικτών. Μήπως θα πρέπει να προσθέσουμε νέες δράσεις στο νέο σχέδιο. Περιμένουμε το έγγραφο για να ξεκινήσει η συνεργασία μεταξύ των πολιτικών ομάδων και να συνεργαστούμε προκειμένου να υλοποιήσουμε τους στόχους και του προηγούμενο σχεδίου δράσης. Ευχαριστούμε κυρία Γκαρσία Πέρεση, κυρία Ράς. Ευχαριστώ. Σίγουρα τα ζώα είναι σύντροφοι του ανθρώπου, ε, είναι τρόφιμο, μερικές φορές γίνονται τρόφιμο, χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή κάποιων γεωργικών εργασιών Ασχοληθήκαμε με το θέμα των ζώων πολλέ φορέ και στο προηγούμενο κοινοβούλιο και δίκιο έχουν και η κυρία Γέγκλε και η κυρία Πόλσεν. Όταν μιλήσαμε για τη θυσία των ζώων ε, και τη σφαγή τους για να γίνουν τροφή, για τη μεταφορά των ζώων, στις διάφορες ακροάσεις, σεμινάρια και εργαστήρια μελέτης που είχαμε, ακούσαμε πολλούς επιστήμονες που μας είπαν πράγματα που ήταν τελείως άσχετα με τις δικές μας ιδέες, που δεν είχαν καμία σχέση με την εντύπωση που είχαμε εμείς για το θέμα αυτό. Και πολλές φορές η επιστημονική κοινότητα άσκησε κριτική σε επιστημονικές δημοσιεύσεις και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μας μέμφθηκε για αποφάσεις που λάβαμε και που συρίχθηκαν σε προκαταλήψεις μερικές φορές ή σε ιδέες που είχαν, δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Γιατί εμείς δεν είμαστε επιστήμονες, εμείς είμαστε πολιτικοί και εκπρόσωποι των ψηφοφόρων μας. Θα πρέπει όμως να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα και τις εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και τους μηχανισμούς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να καταλήξουμε επιτέλους σε αντικειμενικούς δείκτες της ευημερίας των ζώων. Γιατί πώς θα αξιολογήσουμε ένα σχέδιο δράση σαν αυτό που είχαμε και να το κρίνουμε σωστό ή ακατάλληλο, αν δεν έχουμε επιστημονικές βάσεις. Μπορούμε να έχουμε κάποια εμπειρική γνώση, αλλά άλλο επιστήμη και άλλο εμπειρική γνώση. Χρειαζόμαστε κάποιους αντικειμενικούς δείκτες και έναν ορθολογικό και ισορροπημένο τρόπο εργασίας. Δεν θα πρέπει να μείνουμε στην πρώτη μας σκέψη και στην αισθηκτόδη μας πρόταση, αλλά να λάβουμε υπόψη και κάποια επιστημονικά κριτήρια. Θα πρέπει με βάση τέτοιου αντικειμενικούς επιστημονικούς δείκτες ευημερίας να εκπονήσουμε τις μελλοντικέ μας προτάσεις και αυτές οι προτάσεις να τις εφαρμόσουμε και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αυτό μας ζητούν οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις προστασίας των ζώων. Και ταυτόχρονα θα πρέπει να απαιτήσουμε τέτοιες υψηλές προδιαγραφές και από παραγωγούς τρίτο χωρών που μας στέλνουν, εξάγουν ζώα προς εμάς, γιατί θα πρέπει να πετούμε την ευημερία των ζώων από τη στιγμή της γέννησης μέχρι τη στιγμή της φαγής και όχι σε ορισμένες στιγμές της ζωής τους. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο μεταφορά, μας ενδιαφέρει όλη η διάρκεια της ζωής του ζώου και όλων μας ενδιαφέρουν όλα τα ζώα σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, είτε είναι εντός είτε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό μας ζητούν οι Ευρωπαίοι πολίτες και αυτό απαιτούν και οι ενώσεις προστασίας των ζώων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Ράντς. Η κυρία Μαγκίνες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τα σχόλιά της. Θα ήθελα να κάνω τρία σχόλια πιο συγκεκριμένα αναφέρατε ότι θα πρέπει να υπάρχει να υπάρξει μια νέα οδηγία για, τα, για τη μεταφορά. Ο διάφοροι συνάδελφοι είπαν ότι είναι αφιλεγόμενο αυτό το θέμα. Εγώ ανησυχώ λιγάκι, γιατί το Κοινοβούλιο πάντα ψάχνει για νέες ε, οδηγίες όταν το πρόβλημα είναι στην έλλειψη, ε, στην κακή εφαρμογή των ισχυόντων. Δεν θέλουμε νέο νομοθεσία σε αυτό το τομέα. Ε, στην πραγματικότητα η Κομισιόν και οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να εφαρμόσουν πλήρως την ισχύουσα οδηγία για τις μεταφορές. Αυτό θα πρέπει να προσέξουμε αγαπητοί συναδελφοί, να μην προσθέτουμε νομοθετήματα τα οποία απλώς δεν εφαρμόζονται. Σας παρακαλώ λοιπόν ζητήστε την εφαρμογή των νομοθετημάτων. Αν οι επιθεωρήσει και οι έλεγχοι δεν υπάρχουν, θα πρέπει να μα πει η Κομισιόν σε ποια κρατη δεν υπάρχουν και τι δράσει έχουν ληφθεί, ούτω ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι επιθεωρήσει και οι έλεγχοι λαμβάνουν χώρα. Τώρα, ε, θα ήθελα να σας αναφέρω το θέμα της ε, μεταφοράς των αλόγων. Ε, είναι πολύ ευαίσθητο θέμα. Υπάρχει κόσμος που θέλει και άλλη νομοθεσία, σκληρότερη νομοθεσία. Στην πραγματικότητα δεν εφαρμόζουμε την ισχύουσα νομοθεσία. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ λοιπόν αυτό να λάβετε υπόψη σας. Ε, μου άρεσε το σχόλιο για την επιστημονική απόδειξη και όχι για τα αίσθηκτά μας, έτσι, τις πρώτες μας σκέψεις. Ε, τα σχόλια σας που σας είπαν, που κάνατε για τα αντιβιωτικά, τα άρρωστα ζώα, την υπερβολική χρήση αντιβιωτικών. Ε, ανησυχούν τέτοια σχόλια. Γιατί είναι παράνομο να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και αν σε ορισμένα κράτη-μέλη υπάρχουν υπερβολικά κατάλοιπα, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό από το κράτος μέλος και τις αρμόδιες αρχές του. Νομίζω ότι το δικό μας κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικό στη χρήση των ε, λόγων και λέξεων. Ε, εγώ δεν ε, έχω πληροφορίε για υπερβολική χρήση στη γεωργία, αλλά υπερβολική συνταγογράφηση του, των αντιβιωτικών ε, γενικά στους ανθρώπους. Και αυτό είναι ε, θέμα ανησυχίας. Προσοχή λοιπόν για αυτό το θέμα. Συμμετείχα στην αρχική συζήτηση στο, στην περασμένη κοινοβουλευτική θητεία και νομίζω ότι η εστίαση στα ε, ζώα που εκτρέφονται είναι πολύ σωστή. Εγώ θα ήθελα όμως να εστιάσουμε και σε όλα τα ζώα. Γιατί αν μας ανησυχεί η ευμερία των ζώων, δεν θα πρέπει να περιοριστούμε μόνο σε εκείνα που χρησιμοποιούνται στην διατροφική αλυσίδα. Νομίζω ότι θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας αυτό. Επίσης, προσοχή για, το ότι μόνο η μεγάλη και εντατική γεωργία δημιουργεί προβλήματα. Απλώς δείχνει τα προβλήματα και μπορούμε να τα εντοπίσουμε τα προβλήματα πούμε, ευημερίας πιο έντονα σε αυτή τη γεωργία. Αλλά συχνά η ψυχαγωγική γεωργία δεν, δεν α, προσέχει αρκετά την ευημερία των ζώων. Συχνά ο κόσμος πιστεύει ότι κάνει ό,τι πρέπει, αλλά δεν έχει πραγματικές γνώσεις, τα κτλ. Επομένως είναι ένα ε, τεράστιο ευρύτερο θέμα κοινωνίας. Νομίζω ότι η ευημερία όλων των ζώων είναι σημαντική και αυτό θα πρέπει να προσέξουμε. Ελπίζω λοιπόν να τα καταφέρετε στην ε, προσπάθειά σας. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ την κυρία Μαγκίνες. Ε, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας πω ότι τα προϊόντα φώκιας δημιούργησε ένα τεράστιο προηγούμενο. Απαγορεύσαμε λοιπόν την εισαγωγή τέτοιων προϊόντων ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για λόγους ευημερίας των ζώων. Πιστεύω ότι θα πρέπει να βασιστούμε σε αυτό το προηγούμενο και θα πρέπει να βάλουμε περιορισμούς ε, στην ε, εισαγωγή και στο δικό μας τομέα και σε άλλους τομείς πέρα από τα προϊόντα από φώκες. Όταν τα γεωργικά προϊόντα εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όταν αυτά τα προϊόντα προέρχονται από κτηνοτροφία η οποία δεν ε, σέβεται τους κανόνες τους δικούς μας, αυτές οι εισαγωγές θα πρέπει να απαγορευτούν. Απλούστατα. Όταν πιέζουμε τους ε, γεωργούς μας να χρησιμοποιούν όλο και πιο επιζήμιες μεθόδους, συχνά χάνουν την ανταγωνιστικότητά τους απέναντι σε γεωργούς ε, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που συχνά δεν σέβονται τις ευρωπαϊκές μεθόδους. Να υπενθυμίσω ότι η Ουγγαρία είναι όμορη χώρα της Ουκρανίας. Αν η Ουγγαρία δεν θα τα καταφέρει να παράγει ανταγωνιστικά αυγά, αυγά εξαιτίας της πολύ αυστηρής νομοθεσίας ε, σε ό,τι αφορά το μέγεθος των κλοβών, τα αυγά απλούστατα θα εισαχθούν από μη ευρωπαϊκέ χώρε από την Ουκρανία προκειμένου, στην Ουγγαρία, όπου δεν υπάρχει κανένα απολύτω κανόνα για το περιβάλλον και δεν υπάρχει τίποτα για την προστασία και την ευημερία των ζώων. Θα ήθελα να κάνω ακόμα μια άλλη παρατήρηση. Νομίζω ότι πρέπει να εξετάσουμε όλα τα μέτρα ευημερίας των ζώων και να δούμε τι σχέση έχουμε με την παραγωγικότητα. Εδώ δεν σκέφτομαι μόνο το οικονομικό κέρδος, αλλά το γεγονός ότι τα διάφορα μέτρα για την ευημερία των ζώων προκαλούν μία αύξηση της ποσότητας των ζωοτροφών. Μην ξεχνάτε ότι ένα επιπλέον τόνος ζωοτροφών προϋποθέτει ένα κυβικό μέτρο επιπλέον νερού. Με αυτά τα μέτρα λοιπόν προκαλούμε την διασπάθηση εκατομμυρίων κυβικών ε, ε, μέτρων νερού και απορρίψεων επίση καταλήπων στο περιβάλλον. Μην ξεχνάτε λοιπόν και την περιβαλλοντική διάσταση του πράγματος. Ευχαριστώ. Ο κύριο Άγνιου. Ευχαριστώ ε, για τις αθέλητες συνέπειες ε, της θετικής νομοθεσίας για την ευημερία των ζώων. Καταρχάς, α, τους κλωβούς για τους οποίους μίλησε ο Ούγγρος συνάδελφος. ελπίζω να γνωρίζει η Επιτροπή ότι η θνησιμότητα στα, στους κλοβούς είναι πολύ μικρότερη από την, μορτάλ, από την ε, θνησιμότητα συγγνώμη, των πουλερικών α, ελεύθερης, ελεύθερης βοσκής. Παραδείγματο χάρη, ε, τα πουλερικά ελεύθερης βοσκής, ας πούμε, επιτίθενται σε, δέχονται μάλλον επιθέτησης από άλλα ζώα και απλώς θα τα σκοτώνουν. Συχνά, α πούμε, ένα πτηνό, παραδείγματο χάρη, έρχεται, το χτυπάει το πουλερικό στο, στο κεφάλι, ε, παθαίνει ασφυξία ή το, το ραμφίζει πολύ έντονα. Καταλαβαίνετε αυτοί, αυτές είναι οι συνέπειες, οι κακές από την καλή νομοθεσία. Ακούσαμε ήδη τον Ούγκρο συνάδελφο που μίλησε για το πρόβλημα με τους κλωβούς. Συμφωνώ απόλυτα με τα σχόλιά του. Αν ε, τα μέτρα αυτά προχωρήσουν ε, την 1η Ιανουαρίου 2012, θα εισαγάγουμε τελικά προϊόντα σε μεγάλες ποσότητες από το εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακαλώ να το ξανασκεφτούμε και να επιβάλλουμε μία καθυστέρηση. Ε, να έχουμε κάποια διαρθρωμένα μέτρα, ούτω ώστε να έχει η βιομηχανία περισσότερο χρόνο να προσαρμοστεί για το θέμα αυτό των κλοβών. José Euh, euh, euh, Ευχαριστώ. Λέει ο κύριος Μποβέ. Ένα προήμιο. Συμφωνώ και καταλαβαίνω τις ε, προθέσεις της κυρίας ε, Πόλσεν. Να υπενθυμίσω όμως το εξής. Είμαστε εδώ πέρα για να εκτρέψουμε ζώα και όχι για να παράγουμε κρέας. Αυτή είναι μια άλλη σχέση με το ζώο, αν είμαστε εκτροφείς και όχι παραγωγή κρέατος, έτσι. Γιατί από τη μία έχουμε τη βιομηχανική σχέση και από την άλλη έχουμε σχέση με τα ζώα. Είναι τελείως διαφορετική αυτή η σχέση. Θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις. Μία πρώτη παρατήρηση για την χρήση των αντιβιωτικών. Δημιουργούν όντω πρόβλημα στα ζώα, αλλά δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα στους γεωργούς και τους μισθωτούς που δουλεύουν ιδίως στα χειροστάσια. Γιατί από την ανάλυση της α, ιατροφαρμακευτικής κάλυψης στη Γαλλία βλέπουμε ότι η ανθεκτικότητα στα αντιβιωτικά ε, στις, στα χειροστάσια ήταν ανάλογη με το μέγεθος του χειροστασίου. Όσο περισσότερα ε, γουρούνια υπήρχαν στο χειροστάσιο, τόσο μεγαλύτερη ήταν η ανθεκτικότητα των αντιβιωτικών ε, η ανθεκτικότητα των στα αντιβιωτικά συγγνώμη, για τους ε, μισθωτούς του χειροστασίου. Επομένως πρέπει να δούμε και τον τρόπο χρήσης ε, των ε, αντιβιωτικών και των φαρμάκων στις ε, εκμεταλλεύσεις. Δεύτερο θέμα. Μιλήσαμε πολύ συχνά για εισαγωγέ. Δεν είναι το θέμα της ανταγωνιστικότητας μεταξύ χωρών, ανταγωνισμού μεταξύ των χωρών που μας απασχολεί, αλλά είναι ο τρόπος μεταξύ με τον οποίο κάποιοι γεωργοί ε, στην Ευρώπη, για να μην σεβαστούν τους κανόνες στην Ευρώπη, πηγαίνουν στη Βραζιλία ή στην Ταϊλάνδη, με μετεγκαθίστανται και εν συνεχεία για να φέρουν τα πουλερικά πίσω στην Ευρώπη ζητάνε και άλλα χρήματα. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Δεν είναι φυσιολογικό. Μια γαλλική επιχείρηση όπως η Ντου που είναι μια μεγάλη εταιρεία να παίρνει επιδοτήσεις για να εξάγει στην Αφρική 60 εκατομμύρια ευρώ πήρε. Και ταυτόχρονα να χρηματοδοτείται πάλι όταν εξάγει από τη Βραζιλία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση κοτόπουλα. Θα πρέπει να γίνουν σεβαστοί οι κανόνες. Είτε είμαστε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ ε, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω την ε, συζήτηση που κάναμε για την ε, εκτροφή βοήου ζώων για βόηο κρέας στη Βραζιλία. Όλα αυτά είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους. Ευχαριστώ. Κύριο Σίνσκακ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολλά από τα επιχειρήματα που ακούσαμε σήμερα θα πρέπει ίσως να ενταχθούν μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Χθες μιλήσαμε για το γαλακτοκομικό τομέα. και το γεγονό ότι συνέχεια στοχεύουμε προ τη μεγαλύτερη παραγωγή. Αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό είναι η αιτία του προβλήματο. Γιατί δημιούργησε μια τεράστια φαρμακοβιομηχανία, α πούμε, για να δίνει φάρμακα στους γεωργού ε, προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγή του γάλακτος. Το ίδιο και εδώ. Τη γνώμη μου αυτό είναι το σημαντικότερο πρόβλημα. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε κάποιες ε, προδιαγραφές ε, υψηλής ποιότητας του γάλακτος για να γνωρίζει ο καταναλωτής ότι ο κτηνοτρόφος ή ο μεταποιητής ε, ε, των χείρων πληρεί κάποιες υψηλές προδιαγραφές και δεν χρησιμοποιεί όλο και περισσότερα αντιβιωτικά στην παραγωγή. Δεν θα πρέπει ε, εμείς οι ίδιοι να συμβάλλουμε στον περιορισμό της διάρκειας ζωής των ζώων. Γιατί έχουμε αποφασίσει σε πόσα χρόνια θα πρέπει να πάει στη σφαγεία η Ελλάδα, αλλά το θέμα είναι στη διάρκεια της ζωής πόσα αντιβιωτικά χρησιμοποιούνται. Το ίδιο και στα χειροστάσια. Τα ίδια προβλήματα υπάρχουν. Δεν είναι μόνο η μεταφορά το πρόβλημα. Η μεταφορά είναι το τελευταίο στάδιο της παραγωγής ε, ε, του κρέατος, για παράδειγμα. Η, της ε, πτυνοτροφίας ή της ε, χειροτροφίας. Το θέμα είναι πριν τη μεταφορά επίσης τι θα συμβεί, γιατί πριν τη μεταφορά είναι που χρησιμοποιούνται τα αντιβιωτικά. Επίσης, υπάρχει το θέμα των κατοικιδίων. Αναφέρθηκε και αυτό. Ίσως θα πρέπει και εκεί να ασχοληθούμε με ευρύτερο θέμα και όχι μόνο με τις μεταφορές. Γιατί πολλές φορές ε, μεταφέρουμε με τα μέσα μεταφοράς κάποια κατοικίδια. Βέβαια δεν είναι πολλά τα κατοικίδια που ταξιδεύουμε το αεροπλάνο. Το θέμα είναι ακόμη και στις καταστάσεις αυτές ε, πώς αναφερόμαστε, πώς ασχολούμαστε με την ευημερία των ζώων. Εγώ δεν έχω προσωπικά κατοικίδιο, αλλά βλέπω πώς ε, οι γείτονέ μου, οι φίλοι μου που ε, τρέφουν τα ζώα τους, ότι τους κάνουν δίαιτα για παράδειγμα. Κάνουν δίαιτα στο σκύλο τους. Και όταν ε, του δίνουν ένα μπισκότο τροφής, ε, πρέπει να ξέρουν τι ακριβώς περιλαμβάνει. Ενώ ο καημένο ο σκύλο, ακριβώ επειδή βρίσκεται στη δίαιτα, περνάει τη μέρα πεινασμένο, περιμένοντα το επόμενο μπισκοτάκι. Τέτοιου είδου καταστάσει ε, εκτιλήσονται μπροστά στα μάτια μα. Θα πρέπει λοιπόν και αυτά τα θέματα να τα λάβουμε υπόψη. Ο κύριο Ποιος... Δεν είναι μόνο τα ζώα που υποφέρουν από τις δίαιτες και άνθρωποι υποφέρουν, αλλά τι να κάνουμε, αυτά έχει ζωή. Θα ήθελα να πω στο συμπατριώτη μου ότι ο Τσέσοφ και όντως κάνει, κάνει αλλά μόνο σε τις επιβάλλει, δεν του επιβάλλει κάποιος άλλο ενώ στα ζώα υφίστανται τις δίαιτες χωρίς να τις διαλέγουν. Έχουμε υψηλέ προδιαγραφέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ευημερία των ζώων και πολύ ωραία. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Είναι τιμή μας και δείχνει το, την υψηλή ανάπτυξη και τον υψηλό πολιτισμό της κοινωνίας μας. Οι ψηλέ προδιαγραφές όμω ε, αυξάνουν και τι δαπάνε, αυξάνουν το κόστος της γεωργικής μας παραγωγής. Και έτσι η γεωργική παραγωγή γίνεται, ε, δεν ε, γίνεται, μη προσοδοφόρα. Χάνει τα περιθώρια κέρδους. Και όχι μόνο αυτό, ακόμη και οι ζημιές έχουν οι γεωργοί μας. όταν δεν πληρούν αυτές τις ψηλές προδιαγραφές. Και πολλές φορές η διοίκηση, η γραφειοκρατία και εμείς υποχρεώνουμε στην ε, τήρηση των υψηλών προδιαγραφών της δικής μας παραγωγής, αλλά θα πρέπει να το εφαρμόζουμε και για τα εισαγόμενα προϊόντα. Γιατί αν υπάρχουν ζημίες ε, για τους δικούς μας γεωργούς, θα πρέπει να αντισταθμίζονται. Και εμείς είμαστε υπεύθυνοι απέναντι στους παραγωγούς μας. Έχουμε να δώσουμε λόγο απέναντι στους. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε αυτό το θέμα και στις διαπραγματεύσεις με την Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου. Και οι διαπραγματευτές μας εκεί να μας ενημερώνουν για το πώς ε, εκτελήσονται οι διαπραγματεύσεις στην Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου. Ευχαριστώ. Grazie, onorevole Zegreschi. Un punto molto importante. Mi soffermerò anch'io su questo Σημαντικό σημείο, θα το θίξω και εγώ αργότερα αυτό το σημείο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι το σχέδιο δράσης για την προστασία των ζώων 2006 έως 2010 είναι σωστό και ξεκινήσαμε με βάση το πρόγραμμα αυτό πολλές συζητήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίες θα πρέπει να συνεχιστούν. Ιδάλλως, ε, δεν θα υπάρχει συνέχεια στο πρόγραμμα. Μάλλον θα δοθεί εντύπωση ότι απότομα διακόπη. Κατά δεύτερον, θα πρέπει από τις αποφάσεις που λάβαμε στο πρωτοσχέδιο αντράσεις να αφαιρεθούν κάποια θέματα. Καταρχάς η γραφειοκρατία, να προσέχουμε να μην δημιουργούμε με τις ίδιες μας τις ρυθμίσεις γραφειοκρατία στις ε, χώρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Το δεύτερο που ήθελα να παρακαλέσω την κυρία Πάουλσεν και με ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι ο βαθμός εφαρμογής στα διάφορα κράτη-μέλη, γιατί δεν έχει νόημα να δημιουργούμε νέα προγράμματα και να μένουν περιφέρειες ή κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να εστερούν και αυτό θα αποτελέσει, αν θέλετε, αποτρεπτικό παράγοντα και για άλλες χώρες. Το τρίτο θέμα που αναφέρθηκε επίσης πολλές φορές σε ό,τι αφορά την εξωτερική προστασία. Το είπαν και οι δύο συνάδελφοι δεν μπορεί να διαιρεθεί η προστασία των ζώων. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε πρότυπα τα οποία θεωρούμε απαραίτητα και σωστά και εύλογα. Και παράλληλα να μην ισχύουν αυτά τα πρότυπα για κάποιες ομάδες ζώων. Θα πρέπει στην διατύπωση να βάλουμε μία δικλίδα ασφαλείας, προκειμένου να μην εξαιρούνται είδη ζώων. να μην ε, είμαστε σαν μικροκυπουροί, να πούμε ότι «Α, κοιτάξτε, εγώ καθάρισα το δικό μου τον κήπο και δεν με νοιάζει τι γίνεται πέρα από το δικό μου τον κήπο». Όχι. Και αυτό θα πρέπει να ισχύσει επί του συνόλου της παραγωγής. Έχουμε αναπτύξει πρότυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να μην επιτρέπουμε τέτοια θέματα. Και αυτό λοιπόν θα πρέπει να συμπεριληφθεί και στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ. Παρακαλώ λοιπόν την ε, εισηγήτρια να το λάβει αυτό υπόψη. Αν το πράξει θα έχει την απόλυτη υποστήριξή μου. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν, στην κυρία Ανδρέα Γκαβινέλη, θα ήθελα να πω και εγώ με τη σειρά μου τι άποψη έχω για αυτό το σημαντικό σημείο. Άκουσα από διάφορους ομιλητές διάφορα πράγματα ε, στρέφουμε λοιπόν προς την κυρία Πόλσεν. Είμαστε περήφανοι που η Ευρώπη έχει νομοθετήματα για την ε, ευημερία των ζώων και μάλιστα τόσο προχωρημένα. Είμαστε σίγουρα περήφανοι γιατί νομίζω ότι για πολλές χώρες του κόσμου αποτελούμε σημείο αναφορά. Παρ' όλα αυτά, όπως υπόθηκε και προηγουμένως, γνωρίζουμε ότι υπάρχει κίνδυνος αθέμητου ανταγωνισμού ή στρέβλωση του ανταγωνισμού, αν προτιμάτε, για τους παραγωγούς μας ε, απέναντι σε άλλες ε, χώρες, γιατί άλλες χώρες δεν ακολουθούν τους ίδιους κανόνες, αλλά έχουν ελεύθερη πρόσβαση με, για τα προϊόντα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, για αυτό το θέμα των πουλερικών, ας πούμε, είναι θέμα πασιφανές οι παραγωγοί που εξάγουν στην Ευρώπη θα πρέπει να σέβονται τους ίδιους κανόνες ευημερία των ζώων. Αν δεν το κάνουμε αυτό, απλώς μετεγκαθιστούμε τις εκμεταλλεύσεις εκεί που οι κανόνες δεν υπάρχουν. Νομίζω ότι στο, στην πολυμερή τράπεζα του ΠΟΕ θα πρέπει όχι απλώς να είμαστε οι πρώτοι στην τάξη για τα, τους κανόνες ε, ευημερίας των ζώων, αλλά θα πρέπει να κάνουμε και τις άλλες χώρες να σεβαστούν αυτούς τους κανόνες, οι οποίες εν συνεχεία εξάγουν τα προϊόντα τους στην Ευρώπη. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό και τονίστηκε και θα ήθελα και εγώ να το υπογραμμίσω. Αντρέα Γκαβινέλη, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχετε το λόγο. Α, συγγνώμη, ο Άλμπερντ Ντες πρώτα. Ε, ζήτησε το λόγο, δεν σα είχα δει, Άλμπερτ, συγγνώμη. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ζήτησα το λόγο στην ε, αρχή, αλλά δεν πειράζει να τον πάρω τώρα το λόγο. Θα ήθελα να τονίσω πολλά από αυτά που ακούσαμε. Οι απαιτήσει αυτές είναι εύλογες, αλλά τα έθιξε αυτά και ο Πρόεδρος. Θα πρέπει να προσέξουμε και στο σημείο αυτό και αυτά που αναφέραμε για την έρευνα, να μην μετακατασταθούν τμήματα της έρευνας εκτός Ευρώπης, στην Βραζιλία, στην Λατινική Αμερική, γιατί προεθούμε, για παράδειγμα, κλιματιζόμενα φορτηγά και εκεί με 40 βαθμούς Κελσίου δεν έχουν καν ε, κλιματισμό στα φορτηγά. Δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Να μην το επιτρέψουμε. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό και στους εκτροφείς ε, και σε όλο τον κόσμο εδώ στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να τον υπορφορτώσουμε με ρυθμίσεις. Να πω όμως και δύο λόγια για τα αντιβιωτικά. Θα πρέπει να το συζητήσουμε με μεγάλη προσοχή γιατί και στο Γερμανικό Κοινοβούλιο πήρε χρόνο η συζήτηση αυτή χωρίς... Ε, υπάρχουν μάλλον επιστημονικά στοιχεία που καταδεικνύουν ότι η χρήση αντιβιωτικών είναι η πιο υψηλή, πιο υψηλή από κάθε άλλο είδος στα πουλερικά εκτροφής. Και κοιτώντας και τα ποσοστά θνησιμότητας, ε, διαπιστώθηκε ότι σε κλωβούς ε, το ποσοστό θνησιμότητας είναι 6% και σε πουλερικά ελεύθερης εκτροφής 12 15% και ένας συνάδελφος είχε επισημάνει ότι η μητέρα του που είχε ε, κοτόπουλα ήταν 100% το ποσοστό θνησιμότητας επειδή κυκλοφορούσαν λεπούδες. Άρα θα πρέπει να θέσουμε σωστές προτεραιότητες. Αναφέρθηκαν και τα εικόσιτα ζώα. Όταν επιστρέφω στο σπίτι μου και έχω ένα πολύ όμορφο retriever, golden retriever, τριών χρονών. Όταν κάθεται στον καναπέ και μαγειρεύω διάφορες βαβαρικές σπεσιαλιτές και έρχεται δίπλα μου και στέκεται. Και του λέω, τι κοίταξε Ρίκο, έχω τύψεις που σε βλέπω, γιατί τα περνάς καλύτερα από ότι εκατομμύρια άνθρωποι σε αυτόν τον πλανήτη. Έχεις καναπέ, φαγητό, νερό, ελευθερία, παίζεις κάθε μέρα. Θα πρέπει λοιπόν να ξέρουμε ότι υπάρχουν δισεκατομμύρια άνθρωποι που περνούν χειρότερα από ό,τι τα ζώα μας συνήθως. Και θα πρέπει λοιπόν να θέσουμε σωστές προτεραιότητες, να είναι σταθμισμένη, ισορροπημένη η προστασία των ζώων που θα περάσει, όχι για να καθησυχάσουμε απλά τις τύψεις μας. Ήταν τεράστιες οι συζητήσεις. Ε, στη Γερμανία για τις μεταφορές τροφίμων στο Λίβανο. Τερματίστηκαν. σήμερα μεταφέρονται οι... τα προϊόντα αυτά από, το... από την Βραζιλία και από άλλες χώρες. Κέρδισε κάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα πρέπει να το διευκρινίσουμε. Είμαι πεπισμένος ότι οι δικέ μα μεταφορέ ζώων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πολύ καλύτερε από αυτέ που γίνονται σήμερα. Άρα δεν έχει νόημα να καθησυχάζουμε τι δικέ μα τι τύψει και τελικά αυτό να αποβαίνει βάρο άλλων ζώων αλλού στον πλανήτη. Ευχαριστώ. Είμαστε πεπισμένοι ότι το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και όλοι θα πρέπει να ασχοληθούμε, όλοι θα πρέπει να εμπλακούμε. Ευχαριστώ. Πριν ξαναδώσω, πριν δώσω μάλλον ξαναδώσω το λόγο στην κυρία Πόλσεν, ας δώσω επιτέλους το λόγο ε, στον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Ο κύριος Γκαβινέλη. Ευχαριστώ κύριε Ντεκάστρο. Καλημέρα σε όλα τα μέλη τη Επιτροπή και θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Πόλσον εν ονόμα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτή την έκθεση πρωτοβουλία. Είμαι ο υπεύθυνο αυτού του τομέα, όπω είπατε. Εδώ και αρκετό καιρό ασχολούμαι με την προστασία των ζώων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 15 χρόνια ασχολούμαι με αυτό το θέμα. Θα ήθελα να σα πω ότι δεν υπάρχει καταλληλότερη χρονική στιγμή από αυτή τη σημερινή για να μιλήσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ένα τέτοιο θέμα, για να υπάρξει μια τέτοια έκθεση πρωτοβουλία. Αυτό που άλλαξε σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση είναι το μελλοντικό σχέδιο δράσης. Κατά την άποψη της Επιτροπή, θα υπάρξει μια ευαίσθητη αλλαγή σε ό,τι αφορά την ε, ευθύνη των ε, οργάνων της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στους πολίτες σε αυτό το τομέα. Με τη νέα συνθήκη ορίζεται ο, ορίζονται τα ζώα ως ε, όντα που αισθάνονται σε ένα άρθρο της συνθήκης. Και υπάρχει ένα καθεστώς συναπόφασης για οποιοδήποτε τομέα αφορά την προστασία των ζώων. Ενώ μέχρι τούδε είχαμε απλώς μία σχέση διαβούλευσης. Επομένως, το θέμα της α, θέσης, της τάσης των πολιτών δεν έχει, δεν έχει αλλάξει. Επίσης, το θέμα των οικόστων ζώων το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Ε, είτε οι κόστα ζώα αυτά είναι που ζουν κανονικά με στο σπίτι, είτε είναι κότες, που παράγουν ε, αυγά θεωρούνται ε, ζώα που αισθάνονται με βάση τη συνθήκη. Το γνωρίζει λοιπόν αυτό η Κομισιόν. Γι' αυτό το σχέδιο δράσεως του 2006 ε, προέβλεψε επενδύσεις. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες δράσεις. Υπάρχει το welfare quality είναι το πιο μεγάλο πρόγραμμα παγκόσμιας εμβέλειας σε αυτόν τον τομέα, όπου υπήρξε συνεργασία σε διεθνές επίπεδο ε, επιστημόνων και με πολλούς άλλους εμπορικούς εταίρους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι η ευημερία των ζώων ε, γίνεται σεβαστή, αλλά όχι με άκαμπτα μέτρα και πρότυπα για την εκτροφή, αλλά με μέτρα που θέτουν στο κέντρο του το ίδιο το ζώο με βάση συγκεκριμένους δείκτες για το ζώο και για την κατάστασή του. Ε, επίσης θα πρέπει να εντάξουμε την ευημερία των ζώων στη γεωργία και στις γεωργικές πολιτικές. Και πρόκειται για μια έννοια ποιότητα. Γι' αυτό η Κομισιόν εδώ και λίγες μέρες έχει υιοθετήσει μια έκθεση για την επισήμανση της ευημερίας των ζώων που έχει σταλεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια έκθεση η οποία βασίζεται σε ε, μια μελέτη σκοπιμότητας μετά από μια διαβούλευση με πάνω από 110 ενδιαφερόμενα μέρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτροφείς, πολίτες, καταναλωτές, ε, εταιρείε ευημερία των ζώων κτλ. Να μην ξεχνάμε και τις εμπορικές πτυχές όμως ε, σε αυτή την ε, έκθεση επισήμασης και στη σχέση μας με τις τρίτες χώρες. Θα θέλαμε να θέσουμε την ευημερία των ζώων στο κέντρο αυτής της προσπάθειας. Ε, με χώρες όπως η Χιλή, ο Καναδάς, σε διμερές επίπεδο έχουμε προβεί σε διάφορα μέτρα. Έχουμε συνεργασία με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία και θα υπογράψουμε τέτοια συμφωνία με την Κορέα, ε, πάλι για την ευμερία των ζώων, πάντα σε διμερές επίπεδο. Ε, με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε μια διαβούλευση και ένα σχέδιο δράσης τα επόμενα χρόνια. Οι εμπορικοί εταίροι τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καταλάβουν προ τα πού κινείται το μέλλον. Οι γραμμέ ε, είναι πάρα πολλέ. Τι ανέφερα. Κλείνοντα, θέλω να σα πω ότι η Κομισιόν είναι σε μια μεταβατική φάση, πολύ σημαντική. Δεν έχει τίποτα αποφασιστεί οριστικά σε ό,τι αφορά αυτό το πολύ ευρύ και δύσκολο θέμα για τα επόμενα πέντε χρόνια. Και είναι λοιπόν η κατάλληλη χρονική στιγμή για να στραφούμε προς πολιτικές που θέτουν στο κέντρο τους τον, Ευρωπα... τον Ευρωπαίο πολίτη, που ζητάνε απαντήσεις. Συχνά είναι κατεπίγουσες οι απαντήσεις, όπως παραδείγματο χάρη την κλωνοποίηση των ζώων και που θέτουν πάρα πολλά ερωτήματα τα οποία ζητάνε εκατομμύρια πολίτες. Αν γίνει μια τέτοια πρωτοβουλία όπως αυτή ε, η πρωτοβουλία των πολιτών που αναφέρει η νέα συνθήκη. Να μην ξεχνάτε ότι αυτό είναι ένα τομέα ε, όπου τα μάτια των ε, πολιτών στρέφονται. Λαμβάνουμε εκατοντάδες χιλιάδες mail για το θέμα αυτό. Είτε πρόκειται για κότα, είτε για χιμπατζή, είτε για οτιδήποτε για πίθηκο ας πούμε, οι πολίτες θέλουν απαντήσει Ευχαριστώ τον Ανδρέα Γκαπιντέλη. Κυρία Γέγκλε, θα ήθελε να κάνει συγκεκριμένο ερώτημα. Αξιότιμη κυρία Γκαμπινέλη, θυμάμαι στη συζήτηση για το σχέδιο δράσης το 2005 ότι είχατε πει ότι χρειαζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση υψηλά πρότυπα για την προστασία των ζώων σε ό,τι αφορά τα ζώα εκτροφής γιατί ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είμαστε φωτεινό παράδειγμα για όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Και είχατε πει ότι παγκοσμίω οι πολίτες αναμένουν υψηλά πρότυπα από εμάς αναφορικά με τα άλλα κράτη παγκοσμίω. Και αναφέρατε κάποια παραδείγματα. Δεν έχω ε, χρόνο για να τα αναφέρω, αλλά θα μπορούσατε ίσως γραπτά να μας πείτε να μας απαντήσετε για τι ποσότητες μιλάμε. Δεν θίξατε για παράδειγμα τη Βραζιλία και άλλες σημαντικές χώρες. Για τι ποσοστά, τι όγκο μιλάμε και σε ποιο βαθμό επέτρεσε πραγματικά αυτό το φωτεινό παράδειγμα το οποίο θέσαμε. Τι αποτελέσματα υπήρξαν δηλαδή. Κύριος Γκαβινέλη, ευχαριστώ Πρόεδρε. Για τη συζήτηση θα μπορούσα να σας χορηγήσω εξ ονόματος της Κομισιόν ένα σημείωμα με τις λεπτομέρειες και όλες τις εξελίξεις στο, σε διεθνές πεδίο που θα μπορούσε να βοηθήσει την συζήτηση. Παραδείγματο χάρη έχουμε πετύχει αποτελέσματα. Η Διεθνής Οργάνωση για την Υγεία των Ζώων έχει υιοθετήσει το 2006 τα διεθνή πρότυπα για την προστασία των ζώων και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους και τη στιγμή της φαγής τους. Ε, επίσης ε, προβλέπουμε ε, τον έλεγχο των μολυσματικών ασθενειών. Κατευθυντήριες γραμμές επίσης ε, για τον έλεγχο των σκύλων που έχουν λύσα. Είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να ελέγξουμε και την λύσα στις αντισώμενες χώρες. Ε, δέχομαι πολύ καλά αυτό. Δέχομαι πολύ αυτό που μου ζητάτε και μπορώ να σας, έχω, μπορώ να σας δώσω, εξασφαλίσω και διμερείς έτσι, επαφές, προσωπικές επαφές για να σας δώσω και άλλες απαντήσεις. Λοιπόν, κυρία Πόλσεν, και συνεχεία θα περάσουμε στο επόμενο σημείο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ ε, ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Και στη συζήτηση ανακύπτει ότι όλοι έχουμε τις ίδιες ανησυχίες. Αναρωτιέμαι αν η συζήτηση αυτή για την προστασία των ζώων περιλαμβάνει πολλά και διαφορετικά θέματα, πολλές και διαφορετικές πτυχές. και πλέον ε, νομίζω ότι έχει βελτιωθεί πολύ η κατάσταση σε σχέση με το παρελθόν, γιατί περιλαμβάνονται και πολλά θέματα. Για παράδειγμα, τα αντιβιωτικά. Τα αντιβιωτικά δεν μπορεί να χρησιμοποιούνται προληπτικά για να προλαμβάνονται ασθένειες. Και δεν υπάρχει κανένας έλεγχος ουσιαστικά για την ποσότητα των αντιβιωτικών που καταναλώνονται. Δεν ξέρω δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να μου δοθεί μια απάντηση στο ερώτημα αυτό, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ ουσιώδες το θέμα. Πώς ε, ελέγχονται, πώς ε, προστατεύονται τα ζώα. Υπάρχουν συστήματα τα οποία ισχύουν ιδιαίτερα για τους ε, χείρους, για τα πουλερικά, τα οποία προσλαμβάνουν ημερησίως αντιβιωτικά. Ναι, μεν έχει νόημα να χορηγούνται αντιβιωτικά σε ε, ζώα που πάσχουν από ασθένειες, αλλά όχι προληπτικά. Γιατί αλλιώς τίθονται θέματα α, αντοχής στα αντιβιωτικά. Στις κάτω χώρες είναι πολύ περιοριστική η ρύθμιση για τη χορήγηση αντιβιωτικών και για τους ανθρώπους, αλλά δεν υπάρχει κανένας περιορισμό σε ό,τι αφορά τα ζώα. Για παράδειγμα, τα πουλερικά, τους χείρους. Και διαπιστώνουμε ότι για τις ε, επιζωοτίες ουσιαστικά αναπτύσσονται υψηλές αντιστάσεις ε, στα αντιβιωτικά στην Σουηδία διενεργήθηκε σχετική μελέτη η οποία και αποκάλυψε ότι είμαστε πολύ περιοριστικοί στην νομοθεσία μας σε ό,τι αφορά τα αντιβιωτικά προς τα ζώα αλλά δεν υπάρχουν περιορισμοί ιδιαίτεροι για τη χορήγηση αντιβιωτικών σε ανθρώπους. Είναι τελείως δηλαδή αντίστροφη η κατάσταση από τις κατοχώρε. Είναι πάρα πολύ σημαντική λοιπόν η συζήτηση αυτά, αυτή και για την προστασία των ε, ζώων. Στη Σουηδία επίσης οι γεωργοί, οι εκτροφείς δεν επιτρέπεται να έχουν ζώα που παράγουν αυγά. Αλλά άλλα μεταποιημένα προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως πρωτήλη τα αυγά αυτά. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε λοιπόν ότι στο σημείο αυτό υπάρχουν και εμπλέκονται και οικονομικοί παράγοντες και αυτός είναι άλλωστε και ο σκοπός σε κάθε περίπτωση Αυτό τι σημαίνει. Ε, φυσικά ένα σύστημα φιλικό προς τα ζώα που προστατεύει τα ζώα είναι πολύ ακριβό. Αλλά όταν τελικά θα θεσπιστεί το σύστημα αυτό ε, είναι πιο αποδοτικό και συνεπάγεται και με καλύτερη ποιότητα στα τρόφιμα, αλλά και είναι και πιο σωστό το σύστημα αυτό για τους εκτροφείς. Άρα λοιπόν, για μας τους πολιτικούς θα πρέπει το θέμα να είναι πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι ο κάθε εκτροφέας έχει τα μέσα που χρειάζεται στη διάθεσή του για να δημιουργήσει και να εφαρμόσει ένα καλό σύστημα. Ίσως με πιο ευνοϊκές πιστώσεις, αλλά αυτό ίσως να μην εμπίπτει στο πεδίο της ε, συζήτησής μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Πόλτσεν. Ας αφήσουμε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα και ας περάσουμε στο δέκατο σημείο της ημέσιας διάταξης, απλοποίηση της ΚΑΠ. Το Μάρτιο του 2009 η Κομισιόν δημοσίευσε μία ανακοίνωση που είναι ένας απολογισμός των δράσεων που ξεκίνησαν από το 2005 και μετά. Όμως το πεδίο εφαρμογή των εργαλείων για να πετύχουμε μια μεγαλύτερη απλούστευση είναι πολύ ευρύ και μπορεί να αφορά καταστάσεις πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Η δική μας Επιτροπή αποφάσισε να κάνει μια έκθεση πρωτοβουλίας με σκοπό να διευκρινίσουμε τέτοια ερωτήματα και να προτείνουμε και κάποιες λύσεις που θα μπορούσαν ε, να εφαρμοστούν και άμεσα από τους γεωργούς. Ο κύριος Ashworth είναι ο εισηγητής αυτής της έκθεσης πρωτοβουλίας και του δίνω με τα χαράς το λόγο. Ο κύριος Ashworth. Uh, um, Ευχαριστώ. Όπως είπατε και στα εισαγωγικά σας σχόλια, το πεδίο εφαρμογή της απλοποίησης της κοινής γεωργικής πολιτικής είναι τεράστιο. Γι' αυτό και έχω πρόβλημα, γιατί πρόκειται για μια έκθεση τη πρωτοβουλία. Και με βάση τους κοινοβουλευτικού κανόνες περιοριζόμαστε αυστηρά και από την άψη τη έκταση και του αριθμού των λέξεων και τη ε, ουσία. Γιατί ναι μεν το πεδίο της συζήτηση είναι ευρύτατο, αλλά η έκταση της έκθεσης ε, είναι περιορισμένη. Πάντως, η δική μου προτεραιότητα είναι η απλοποίηση της κοινή γεωργικής πολιτικής ε, τη στιγμή της εφαρμογή της. Δηλαδή, θα πρέπει η κοινή γεωργική πολιτική να είναι απλούστερη στην ερμηνεία και πιο προσιτή για το γεωργό και τις γεωργικές επιχειρήσεις. Σήμερα προβλέπεται η πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Δεν πρόκειται να επισέλθουμε λοιπόν σε εξονυχιστικές λεπτομέρειες. Θα περιοριστούμε στα γενικά στοιχεία της έκθεσης. Εγώ θα πρέπει να αναζητήσω κάποιους τρόπους για να γίνει πιο προσιτή η απλοποιημένη ΚΑΠ, ε, λιγότερο γραφειοκρατική και άρα να περιοριστεί το κόστος ε, προς τους γεωργούς, το κόστος εφαρμογής της προς τους γεωργούς. Θα επικεντρωθώ σε τρεις άξονες. Καταρχήν θα αναζητήσω κάποια παραδείγματα περί της γραφειοκρατίας υπερβολικής και περιττής καταχρηστικής γραφειοκρατίας προκειμένου να προτείνουμε απλοποίηση και να απαλλάξουμε από αυτό το βάρος τους γεωργούς. Επίσης θα πρέπει να αποφευθεί η επικάλυψη των ελέγχων γιατί πολλές διαδικασίες, ιδιαίτερα στο ελληνικό εμπόριο, περιλαμβάνουν κάποιους ε, κώδικες και προδιαγραφές ανιχνευσιμότητας και πολύ συχνά εφαρμόζονται τα συστήματα αυτά ε, είναι παρόμοια με τα στοιχεία και τους όρους που ζητούν οι, οι κρατικοί φορείς. Θα πρέπει να γίνει ένα είδος εναρμόνισης μεταξύ των διαφόρων προδιαγραφών, ώστε να περιοριστεί ο αριθμός των ελέγχων και σίγουρα να αποφευθεί η επικάλυψη των ελέγχων, η διπλή διεξαγωγή ελέγχων. Και οργανισμοί και ενδιαφερόμενοι τομείς υπέβαλαν Κάποιε προτάσει προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που γνωρίζουν του κανόνε. Για παράδειγμα, μη συμμόρφωση με του κανόνε ω προ την απάτη, ε, παραβίαση κάποιων περιβαλλοντικών ζητημάτων, θεμάτων υγείας καταναλωτή και το καθεξής. Γι' αυτό και χρειάστηκαν κάποιε προκαταρκτικές ε, διαβουλεύσεις με ενώσει γεωργών, συνεταιρισμού και εκπροσώπου ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώ και με τη Σουηδική και τη Δανική ε, με τη Σουηδική Προεδρία και την Ελληνική Κυβέρνηση, γιατί και αυτές ε, θέλουν να προτείνουν τρόπους απλούστευση τη ΚΑΠ. Η Επιτροπή μας έχει μία μοναδική ευκαιρία να προωθήσει μία, μία έκθεση που θα ε, ελαφρύνει το βάρος της γραφειοκρατίας για τους γεωργούς και θα κάνει την κοινή γεωργική πολιτική πιο φιλική προς το γεωργό. Γι' αυτό και περιμένω τις ε, συστάσεις και προτάσεις των μελών της Επιτροπής. Θα έχω και κατηδία συνομιλίες ε, με τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας, αλλά και με τις πολιτικές τους ομάδες, προκειμένου να επιτύχουμε μια υπερκομματική συνένεση για την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ τον κύριο Ashworth και τώρα ξεκινάει η συζήτηση. Ε, ήδη κάποιοι ζήτησαν το λόγο. Σας υπενθυμίζω ότι έχουμε κι άλλο σημείο στη μέση διάταξη, ένα-δύο σημεία μάλιστα πριν κλείσουμε την ε, πρωινή μας συνεδρίαση. Θα δώσω πάρα αυτό το λόγο στον κύριο Λαβία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας, γιατί μας επιτρέπει να ασχοληθούμε με ένα θέμα που είναι πάρα πολύ προβληματικό για τις γεωργικές μας εκμεταλλεύσεις και τους ε, και τον κλάδο. αυτή τη ΚΑΠ σημαίνει μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα στι γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Γιατί όσο λιγότερο χρόνο ε, σπαταλάτε στι διοικητικέ ε, δουλειέ και στη γραφειοκρατία, τόσο περισσότερο χρόνο μένει για τι παραγωγικέ δραστηριότητε. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, βοηθάμε τις επιχειρήσεις για να είναι ανταγωνιστικέ. Συμφωνώ με τι κατευθυντριές γραμμέ που μα παρουσίασε ο εισηγητή. Πέρα όμω από εκείνο που προβλέπετε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωσή της και στα ζητήματα που ανέφερε ε, ως ζητήματα που προωθούν την απλούστευση, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε περαιτέρω διευκρινήσεις. Φυσικά δεν νομίζω ότι αυτό είναι το βήμα ε, στο οποίο έχει νόημα να επισέλθουμε σε λεπτομέρειες. Απλώς θα πρέπει να δώσουμε κάποιες ενδείξεις. Πέρα από αυτά που είπε στην ε, αρχική του παρουσίαση ο εισηγητής. Ναι. Αν έχουμε υπερβολική γραφειοκρατία πρέπει να την ε, καταργήσουμε. Έχουμε επικαλύψεις και αυτό θα πρέπει να σταματήσει. Αλλά θα πρέπει στο σύστημα των άμεσων, ε, των ελέγχων μάλλον των άμεσων επιδοτενδύσεων και ενισχύσεων να μην επαναλαμβάνονται γραφειοκρατικοί και διοικητικοί έλεγχοι ε, τόσο επιτόπου όσο και βάση εγγράφων αυτοί, αυτές οι επικαλύψεις θα πρέπει να σταματήσουν. Επίσης θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ένα άλλο θέμα που συνδέεται με αυτό που θα συζητήσουμε σήμερα το απόγευμα όταν μιλήσουμε για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ μετά το 2013. Είναι σαφές ότι τα δύο θέματα θα πρέπει να τα συνδυάσουμε και να προβλέψουμε μια νέα γεωργική πολιτική η οποία θα είναι λιγότερο γραφειοκρατική, πιο ελεύθερη και όπου το επίπεδο ευαισθητοποίησης ε, και υπευθυνοποίηση των γεωργών θα είναι μεγαλύτερο. Δεν θα πρέπει συνέχεια να υπόκεινται σε ελέγχους. Ε, Επίσης, ε, έγινε μια μελέτη που παρήγγειλε η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας. Εκεί φαίνεται ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ των διαφόρων χωρών που δεν οφείλονται μόνο στις διαρθωτικές αλλαγές των γεωργικών εκμεταλλεύσεων των επιμέρους κρατών μελών, αλλά και σε διάφορα συστήματα που έχουν αναπτυχθεί εκ παραλλήλου στην, στην κάθε χώρα για να υποστηριχθούν οι γεωργοί. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε και μια τέτοια προσπάθεια για να διαδώσουμε τις καλύτερες πρακτικές, τις βέλτιστες πρακτικές, ούτως ώστε να μειωθούν τα διοικητικά άχθη για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Ευχαριστώ. Η κυρία Κλάς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή που με την ε, έκθεση πρωτοβουλίας του θίγει και κάποια ζητήματα για την απλούστευση της ε, ΚΑΠ. Δεν θα μπούμε κατευθείαν σε λεπτομέρειες, αλλά δεν μπορώ να μιλάω έτσι γενικά για την ε, μείωση της γραφειοκρατίας. Το συζητάμε εδώ και δεκαετίες το θέμα αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να είμαστε σε πιο συγκεκριμένοι. Την τελευταία θητεία συζητήσαμε διάφορα θέματα και είπαμε ότι θέλουμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις ευρωπαϊκές, ε, τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς από κοινού και μετά να υπάρχει και ο κανονισμός για τον ίνο και θεωρήσαμε ότι ήταν μεγάλο στοιχείο για την αφαίρεση της γραφειοκρατίας ε, το στοιχείο αυτό. Αλλά τότε είχαμε μία απαστράπτουσα ιδέα. Είχαμε πει να κοιτάξουμε την ε, οργάνωση της αγοράς του ίνου και αν υπάρχουν τεχνικές ε, λεπτομέρειες, τεχνικοί όροι, να το εξετάσει αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ίσως όλες οι αρμοδιότητες ε, στην οργάνωση της αγοράς να εξαβρεθούν και για τον ίνο. Αυτό θα πρέπει να ήταν τεχνικώς ε, εφικτό. Το έχει υποσχεθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν το εφήρμοσε όμως. Θα ήθελα λοιπόν να το ξαναθέξουμε το θέμα αυτό. Και μιλώ μόνο για τον ίνο, όταν μιλάμε για τα σιτηρά, για το γάλα. Να υπάρχουν όλα τα ρυθμιστικά στοιχεία. Νομίζω ότι αυτό θα αποτελούσε ένα καλό βήμα προς την ε, απλοποίηση. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα νέα μέσα επικοινωνίας για τις ε, πιο αυστηρούς, πιο συχνούς ελέγχους. Και εδώ θα πρέπει να καταστρώσουμε μια ευρωπαϊκή πολιτική, να υπάρχουν ίδιοι κανόνες ανταγωνισμού. Αυτό θα πρέπει να προκύψει ως αποτέλεσμα. Και χαίρομαι που επεξεργαζόμαστε το θέμα αυτό στην Επιτροπή μας και ελπίζω ότι θα τεθούν και πολλά συγκεκριμένα ε, παραδείγματα και στην περίπτωση αυτή είμαι αισιόδοξη για το μέλλον της ε, αγροτικής πολιτικής. Κυρία Πατράου Νέβες. Ευχαριστώ. Το θέμα της απλούστευσης και του περιορισμού της γραφειοκρατίας δεν είναι καινούριο. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί πάρα πολλά χρόνια και είναι πολύ σημαντικό. Ήδη από το 2005, τουλάχιστον το 2005, είχαμε ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία απλοποίησης. Συμφωνούμε λοιπόν ότι δεν έχουμε σημειώσει ακόμη εντυπωσιακή πρόοδο. Γι' αυτό και υποχρεωνόμαστε να ασχολούμαστε τακτικά με το θέμα αυτό και να επανερχόμαστε. Σίγουρα η έκθεση αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα στη σωστή κατεύθυνση και γι' αυτό θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή μας. Είναι σημαντικό να γίνει ένα είδος απογραφειοκρατικοποίησης της ΚΑΠ. Προς όφελος κυρίως των γεωργών μας. Γιατί διαπίστωσα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προωθήσει κάποιες πρωτοβουλίες και έχει καταλήξει σε σημαντικά ωφέλη, αλλά αυτά τα ωφέλη τα καρπώνονται οργανώσεις, αλλά δεν πάνε απευθείας στην τσέπη του Γεωργού. Γι' αυτό θα ήθελα να επισημάνω στον εισηγητή μου την ανάγκη η διαδικασία αυτή του περιορισμού της γραφειοκρατίας να ωφελήσει πρώτα απ' όλα τους γεωργούς. Θα έχουμε δύο διαφορετικών ε, ωφέλων. Καταρχήν, ο χρόνος είναι χρήμα, άρα ότι χρόνο εξοικονομήσουν από, την, από τον περιορισμό της γραφειοκρατίας οι γεωργοί είναι προς όφελός τους και μπορούν να τον αφιερώσουν αυτό το χρόνο στην ανάπτυξη της γεωργικής τους δραστηριότητας. Επίσης, πολλοί γεωργοί, ιδιαίτερα από την δική μου πατρίδα, την Πορτογαλία και μάλιστα από τις Αζόρες, επειδή δεν είναι πολύ μορφωμένοι, έχουν πρόβλημα στη συμμόρφωση με τις γραφειοκρατικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι που συρρυκνώνει και τις δυνατότητές τους. Υπάρχουν ευκαιρίες που λόγω της χαμηλής τους μόρφωσης δεν μπορούν να τις εκμεταλλευτούν. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι τοπικοί μηχανισμοί και καλό θα είναι να υπάρχουν και εθνικοί μηχανισμοί εγρήγορσης ώστε να αποφευθούν επιζήμες καταστάσεις για τους γεωργούς συγκεκριμένων ζωνών. Τουλάχιστον να ελαχιστοποιηθούν αυτοί οι κίνδυνοι για τους γεωργούς. Ευχαριστώ. Εστερνιζόμαστε τις αδρές γραμμές της έκθεσης του κυρίου Άσχορθ για την απλοποιημένη ΚΑΠ και αναγνωρίζουμε την ανάγκη επικέντρωσης στις πρακτικές πτυχές εφαρμογής της ΚΑΠ. Θα πρέπει επίσης ε, οι γεωργοί να συνειδητοποιήσουν τα ωφέλη που θα αποκομίσουν από την απλοποίηση της ΚΑΠ. Ταυτόχρονα θα θέλαμε και τα κράτη-μέλη αλλά και οι περιφέρειες να ευαισθητοποιηθούν ε, για τις ανησυχίες αυτές. Έχουμε πολυσύνθετη νομοθεσία που δυστυχώς δεν ευνοεί τη, το να φτάσει η απλοποίηση μέχρι τους Γιώργους. Πολύ συχνά ζητώνται από, τους, από τα εθνικά προγράμματα υποψηφιότητα και ενδιαφέρον, εκδήλωση ενδιαφέροντο από τους γεωργούς, θα ήταν πιο εύκολο να γινόταν κάτι τέτοιο σε τοπικό επίπεδο. Επίσης είναι πολύ δύσκολο μερικές φορές για τον Γεωργό να λάβει ενημέρωση τα κατάλληλα έγγραφα. Γι' αυτό και η προσπάθεια απλούστευσης. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να λάβει υπόψη την ανάγκη να φτάσει αυτή η απλοποίηση όχι μόνο στα κράτη αλλά και στις περιφέρειες και στον τελικό αποδέκτη που είναι ο ίδιος ο Γεωργός. Κύριε Καλινόφσκι, ο κύριος. Ευχαριστώ. Έχω την αίσθηση ότι από τις μέχρι τώρα ενέργειες υπό το σύνθημα της απλοποίησης της ΚΑΠ και της άρσης της περιττής γραφειοκρατίας, αυτό που καταργήσαμε είναι κάποιοι μηχανισμοί ε, της γεωργικής πολιτικής και τον σωστό τρόπο άσκησης της γεωργικής δραστηριότητας. Περιορίστηκαν οι μηχανισμοί παρέμβασης σε κάποιες αγορές, και η συνέχιση των αλλαγών προς την κατεύθυνση αυτή θα αποδυναμώσει την κοινή γεωργική πολιτική. Η άρση των μηχανισμών παρέμβασης στην αγορά τροφίμων θα περιορίσει de facto τη δυνατότητα κάποια σταθεροποίησης της αγοράς και τον περιορισμό του κινδύνου διατάραξης της αγοράς. Το πρόσφατο παράδειγμα και πολύ χαρακτηριστικό ήταν ο γαλακτοκομικό τομέα και οι τιμέ του γάλακτο. Προσοχή λοιπόν. Η διαδικασία απλούστευση τη κοινή γεωργικής πολιτική και των μηχανισμών αυτή τη πολιτική δεν θα πρέπει να οδηγήσει στην απάλληψη του κοινοτικού χαρακτήρα αυτής της πολιτικής. Γιατί αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την σωστή ανάληψη των προκλήσεων της νέας γεωργικής πολιτικής. Γιατί αυτές οι προκλήσεις έχουν συνολικό χαρακτήρα γενικό και θα μπορούσαμε να τις αντιμετωπίσουμε μόνο με κοινού ε, μηχανισμούς που θα έχουν κοινοτική εμβέλεια. Ευχαριστώ. Η κυρία Ράς Γκαρσία. Όντω, εδώ και πολύ καιρό η παραγωγή, που είναι και οι δικαιούχοι των ενισχύσεων τη κοινή γεωργική πολιτική, μα ζητούν επίμονα περιορισμό της γραφειοκρατίας και βελτίωση των διατυπώσεων. Και βέβαια οι τεχνολογικές εξελίξεις ε, πολλαπλασίασαν τις δυνατότητες αυτών των ε, γεωργών και όλοι προτιμούν να έχουν έναν, ε, ένα γραφείο στο οποίο θα πρέπει να αποταθούν. Βέβαια πρέπει να μην γενικεύσουμε αυτή την λογική και να μην την παραμορφώσουμε. Γιατί η εισαγωγή μιας ενιαία κοινή οργάνωση αγοράς ε, ενέχει πολλά προβλήματα. Όπως είπε η κυρία Κλά, καταλήγουμε σε, στην επιδείνωση ορισμένων ε, αγορών που λειτουργούσαν μέχρι στιγμής έβριθμα, όπως στην κόα του ίνου ή του γάλακτος. πολλές φορές ε, ο Γεωργός δεν μπορεί να βρει το κείμενο για την ΚΟΑ και αυτή η απλούστευση είναι όχι μόνο επικίνδυνη αλλά πολλές φορές και επιζήμια για τον πολίτη και ιδιαίτερα για τον Γεωργό. Σε ορισμένους τομείς όπως τα προκυπευτικά υπάρχουν ε, νέες δυνατότητες διανομής αλλά δεν λειτουργούν σωστά και παραπονιούνται οι γεωργοί και οι παραγωγή. Μάλιστα, πολλέ φορέ ε, τα μεγάλα εμπορικά δίκτυα διανομή κάνουν κατάχρηση τη κατάσταση ε, και εκμεταλλεύονται του παραγωγού, οδηγώντα ε, σε πολύ άδικε καταστάσει που τι καταγγέλουν οι παραγωγοί. Προσοχή λοιπόν σε αυτή την προσπάθεια απλοποίηση. Και θα πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία στους παραγωγούς απορροκυβευτικών τη δυνατότητα να προστατευτούν από την καταχρηστική ενέργεια των μεγάλων δικτύων διανομής. Επίσης θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε ό,τι αφορά την διάλυση και την απορρίθμιση κάποιων κοινοτικών κανόνων. Γιατί ίσως ε, γίνει μια απόπειρα επανεθνικοποίησης από ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αρχίσει η κατάρρευση, η κατάργηση των κανόνων και των μηχανισμών. Στην περίπτωση του γάλακτος, πριν από λίγες εβδομάδες χρειάστηκε να επαναχωρήσουμε σε σχέση με ηλιμένες αποφάσεις που ήταν κακές, ακατάλληλες και που ελήφθησαν σε μια ολέθρια χρονική στιγμή. Θα πρέπει λοιπόν να εμποδίσουμε οποιαδήποτε προσπάθεια προλίαση του εδάφους για τη μελλοντική επανεθνικοποίηση τη γεωργικής πολιτική. Και αν συνεχίσουμε αυτές τις απλοποίησεις, όπως μας απειλεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ίσως καταλήξουμε σε μια κατάσταση ακόμη περισσότερων καταχρήσεων και απειλών επανεθνικοποίησης. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αρχίσει να σκέφτεται σοβαρά, τώρα που αλλάζει η σύνθεσή της, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συναπόφευση πολλά θέματα. Πολλά έχουν μείνει εκκρεμή. Ας μην λοιπόν μας δημιουργήσει άλλα μέχρι ότου επιλύσουμε τα ίδια εκκρεμή. Μετά από αυτό το σημείο θα πρέπει να ψηφίσουμε για το προφορικό ερώτημα το οποίο συζητήσαμε σήμερα το πρωί στις συνεδρίες των συντονιστών. Γι' αυτό σας παρακαλώ μην φύγετε. Ο κ. Άλμπερτ ε, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι το 20ο έτος που είμαι βουλευτής. Και δεν θέλω, δεν τολμώ πλέον να λέω ότι θέλω να κάνουμε απλοποίηση, ότι θέλουμε να μειώσουμε την ε, γραφειοκρατία, γιατί δεν μας πιστεύει κανένας. Εύχομαι κάθε επιτυχία στον εισηγητή. Θα μπορούσε να γίνει διάσημος. Θα ήταν ο πρώτος ο οποίος θα πετύχαινε κάτι τέτοιο. Γιατί ως κοινοβούλιο δεν καταφέρνουμε να μειώσουμε καν την γραφειοκρατία εντός του κοινοβουλίου. Συνάδελφοι αγαπητοί, αν αρχίσουν να σας ε, αφηγούμε τι έγινε τους τελευταίους μήνες, τι έζησα με το καθεστώς για τους ε, βοηθούς, δεν θα μας χρόνος, γιατί Κάθε άλλο παρά μείωση της γραφειοκρατίας πετύχαμε. Σημείωσα. Μάλλον θα τα δώσω αυτά τα περιστατικά, τα γεγονότα σε κάποιον κομικό, ο οποίος θα βγάλει ολόκληρο πρόγραμμα. Δεν λέω ότι η Ευρώπη φταίει για όλη την γραφειοκρατία. Μεγάλο μέρος της ευθύνης το φέρουν και τα κρατημέλη και η ίδια Γερμανία. Αλλά έκανα και κάποιες προτάσεις οι οποίες ε, δεν πέρασαν την προηγούμενη φορά γι' αυτό και τις ξαναθέτω εδώ σήμερα. Έχουμε χι αριθμό εκτροφέων στην Ευρώπη. Ξέρουμε ότι τα επόμενα χρόνια 10-15% του, ποσοστού, του ποσού αυτού θα μειωθεί. Αν θέλουμε όντως να μειώσουμε την γραφειοκρατία θα πρέπει να μειωθεί κατά το ίδιο ποσοστό το, ο αριθμός υπαλλήλων στην Γενική Διεύθυνση Γεωργίας στην Επιτροπή. Μόνο αν μειωθεί ο αριθμός αυτός θα καταφέρουμε να μειώσουμε και τη γραφειοκρατία στην Ευρώπη. Ε, Ευχαριστώ. Ε, δυσκολεύεται ο εισηγητής γιατί δεν ε, έχει χώρο για να μιλήσει. Θα ήθελα να μιλήσω μόνο για την ε, οικολογική αιρεσιμότητα. Σε αυτό το τομέα, ξέρω ότι τα πράγματα δεν είναι τα ίδια σε όλα τα κράτη-μέλη, αλλά όταν υπάρχουν πάρα πολλά ε, κριτήρια για αυτό τον τομέα, ο Γεωργός ε, συνήθως, χωρίς να το θέλει, κάνει λάθος. Ε, ενώ η έλεγχη είναι επικοδομητική, όχι πάντα, αλλά συνήθω. Συχνά λοιπόν ο Γιώργο τιμωρείται, ενώ δεν έχει την αίσθηση ότι έχει κάνει κάτι λάθο, γιατί δεν το έχει κάνει συνειδητά. Θα ήθελα πραγματικά να απλουστεύσουμε τα πράγματα σε αυτόν τον τομέα, να έχουμε 4-5 ε, μέτρα ουσιαστικά να εφαρμόζονται παντού, παρά να περιπλέκουμε τα πράγματα γιατί νομίζω με αυτόν τον τρόπο η ζωή, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσει του Γεωργού περιπλέκονται. Θα ήθελα να εστιάσουμε σε αυτόν τον τομέα. Ευχαριστώ, Μάρκ. Μάρτιν Όσλινγκ. Φοβάμαι μόνο ότι θα γίνει πολιτικός αγώνας για την, τον όρο της μείωσης ε, της γραφειοκρατίας. Έχουμε εκπρόσωπο από τη Βαβαρία στην Ευρώπη που είναι υπεύθυνο για θέματα μείωσης γραφειοκρατίας. Αλλά παράλληλα παρέχει, παράγει μεγάλο αριθμό νομολογίας. Πολλά έγγραφα. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσουμε και πιο πολύ τα νέα ηλεκτρονικά μέσα για να μην ξοδεύουμε τόνους χαρτιού, αλλά ξέρω ότι πολλές προδιαγραφές αποσκοπούν στην προστασία και των μικρών επιχειρήσεων. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορώ να πω ότι θα πρέπει να τα καταργήσουμε όλα. Και φυσικά τίθεται και άλλο ένα θέμα σε ό,τι αφορά για τη μείωση της γραφειοκρατίας, γιατί με γίνεται μετεγκατάσταση στις ιδιωτικές ε, επιχειρήσεις, δηλαδή οι εμπορικές επιχειρήσεις θέτουν ε, δικούς τους ελέγχους και έτσι προκύπτει ένα μεγάλο τμήμα της γραφειοκρατίας, το οποίο δεν σχετίζεται με εμά, αλλά με πολιτικές εμπορίες. Βλέπουμε λοιπόν ότι πολλά μεταφέρονται ε, στον ιδιωτικό τομέα, το οποίο στην ε, γεωργία ουσιαστικά συνεπάγεται και υψηλότερο κόστος, δηλαδή υψηλότερο κόστος για τον εκτροφέα. Merci, είναι ρεαλιστικό να πλουστεύσουμε μια πολιτική η οποία πρέπει να λαμβάνει υπόψη πάνω από την πραγματικότητα πάνω ένα, από δύο εκατομμύρια γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Η προηγούμενη πολιτική έδειξε τα όρια της. Όμως η άγουσα της απλούστευσης δεν μας υποχρεώνει να αλλάξουμε εντελώ το σύστημα ατομικής ε, βοήθειας ε, που τέθηκε σε ισχύ πριν από 17-18 χρόνια. Ένας συνάδελφος μίλησε για μέτρα απλούστευσης. Νομίζω ότι σε ό,τι αφορά την αρεσιμότητα, θα πρέπει να έχουμε απλώς την υποχρέωση να υπάρξουν αποτελέσματα. Ε, να μην κοιτάμε μόνο τα μέσα, αλλά τα αποτελέσματα. Ε, γιατί αν λάβουμε υπόψη μας τα τοπικά χαρακτηριστικά ας πούμε, της γεωργίας, συχνά τα αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα. Ε, από την εμπειρία μου εγώ ξέρω ότι κάθε γεωργική εκμετάλλευση είναι ιδιαίτερη περίπτωση. Δεν υπάρχουν δύο γεωργικές εκμεταλλεύσεις που να μοιάζουν. Ε, επειδή λοιπόν προσπαθούμε να λάβουμε υπόψη μας αυτή τη διαφορετική πραγματικότητα, έχουμε όλη αυτή την ατελείωτη χαρτούρα. Ευχαριστώ κύριε Νταντά. Ε, σας ευχαριστώ όλους και τώρα θα ήθελα να ζητήσω από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να συζητήσουμε για την απλούστευση τη ΚΑΠ στο εσωτερικό του Κοινοβουλίου. Είναι μια δραστηριότητα πολύ σημαντική για την Κομισιόν και έχουμε εντατικοποιήσει τις προσπάθειες στην περίοδο 2005-2009. Τώρα όμως πρέπει να στραφούμε προς το μέλλον για να δούμε τι πρέπει να κάνουμε ακόμα. Νομίζω λοιπόν ότι η συνδρομή του Κοινοβουλίου θα μπορούσε να είναι πολύ σημαντική, γιατί μόνη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Χρειάζεται να ακούσει ιδέε και υποδείξει από τα κράτη-μέλη, από του ενδιαφερόμενους, από το Κοινοβούλιο. Ψάχνουμε λοιπόν μονίμως ε, να βρούμε νέε ιδέε, να ακούσουμε νέε ιδέε. Στο μέλλον θα εντατικοποιήσουμε τη σχέση με τους ε, εμπορευόμενους και ένα από τα στοιχεία που υπάρχουν ε, στην ανακοίνωση του Μαρτίου του 2009 είναι ακριβώς αυτό το πρόγραμμα Harvest Experience, ε, δηλαδή εμπειρία της σοδιάς. Ε, με αυτόν τον τρόπο θα, θα ψάξουμε να βρούμε νέες ιδέες για την απλούστευση. Όπως είπαν διάφοροι βουλευτές, δυσκολία της νομοθεσίας δεν οφείλεται μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στην εθνική και περιφερειακή νομοθεσία που υπάρχει. Και εκεί μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Επίσης, θα έρθουμε σε περισσότερη επαφή με τους εκπροσώπους των διαφόρων κρατών μελών. Έχουμε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για την απλούστευση και νομίζω ότι είναι το κατάλληλο βήμα για να ανταλλάξουμε ιδέε για τι βέλτιστες πρακτικέ. Να δούμε τι κάνουμε, τι γίνεται. Γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα που είναι σε αναβρασμό στα κράτη-μέλη, τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να το εφαρμόσουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα είναι σημαντικό για του επόμενου μήνε και χρόνια. Περιμένουμε λοιπόν με αρκετό ενδιαφέρον το περιεχόμενο της εκθεσής σας και προφανώς θα σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε μελλοντική μας δράση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Αν συμφωνείτε, ας αφήσουμε αυτό το σημείο και ας περάσουμε πάρα αυτά. Θέλετε να πάρετε το λόγο, κύριε Άσχουρθ. Ο εισηγητής, βεβαίως, να δώσουμε το λόγο στον εισηγητή. Ε, σύντομα, δύο λόγια, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις ε, ιδέες του και την συνδρομή τους. Σημείωσα ότι υπάρχει μια προσδοκία ή μια επιθυμία να μειωθεί η γραφειοκρατία, αλλά υπάρχει και μια αίσθηση ότι όλα αυτά τα έχουμε ξανακούσει. Θέλω να καθησυχάσω τους συναδέλφους, ε, γιατί πιστεύω ότι μπορούμε να, να πετύχουμε πράγματα, αλλά να τους υπενθυμίσω ότι δεν είναι η δική μου εντολή να επανεφεύρω τον, την ΚΑΠ. Έτσι. Ίσως αυτό έρθει αργότερα, ε, το 2013. Η δική μου δουλειά είναι η απλούστευση. Να κοιτάξουμε συγκεκριμένες λίγες σε αριθμό περιοχές όπου εκεί μπορούμε να προχωρήσουμε. Ακούγοντας τους συναδέλφου, εντόπισα τρεις τομεί που έρχονται και επανέρχονται στις παρεμβάσεις. Πρώτον, η πρόσβαση, η προσπελασιμότητα της ΚΑΠ. πρόσβαση στον, στο ίντερνετ, τις νομοθεσίες για την ΚΟΑ, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι, πρέπει να είναι απλή η ΚΑΠ, ε, γιατί είναι αυτό σημαντικό για να μπορούν να εφαρμόσουν τους κανόνες οι γεωργοί. Επίσης, πολλοί έχουν την άποψη ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι παραμένει κοινή α, γεωργική πολιτική σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, οι τοπικές οι εθνικές ερμηνείες μοιάζει να είναι πρόβλημα. Και πρέπει να υπάρχει κοινοποίηση των βέλτιστων πρακτικών. Πρέπει να το εξετάσουμε αυτό το τομέα. Επαναλαμβάνω όμως ότι ευχαριστώ τους συναδέλφους, τους ενθαρρύνω να μου δώσουν οποιαδήποτε ιδέα έχουν, ούτω ώστε να ολοκληρώσουμε αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ, κύριε Ashworth. Πολύ ωραία δουλειά. Προχωράμε και με αυτό το δύσκολο και ευαίσθητο θέμα. Ας ε, προσπεράσουμε το σημείο 11 και ας περάσουμε στην προφορική ερώτηση. Σήμερα το πρωί με τους συντονιστές ξεκινήσαμε αυτή τη συζήτηση και καταλήξαμε ότι έχει νόημα να υποβάλουμε αυτό το προφορικό ερώτημα προς την Κομισιόν. Για αυτό το non-paper που έχει εκδώσει η Επιτροπή και που αφορά την ε, μεταρρύθμιση του απολογισμός, λέγεται απολογισμός, αλλάζουμε την Ευρώπη. Έχουμε ετοιμάσει ένα κείμενο μιας σελίδας με συγκεκριμένες ερωτήσεις προς την Κομισιόν και νομίζω ότι θα πρέπει να ψηφίσουμε αυτό το κείμενο, γιατί αν ε, συμφωνείτε μπορούμε να το δρομολογήσουμε το θέμα. Ελπίζω να κοιτάξατε αυτό το σχέδιο κειμένου και αν συμφωνείτε θα πρέπει επίσημα να θέσω σε ψηφοφορία αυτό το κείμενο. Σας ρωτώ, συμφωνείτε ποιος είναι υπέρ του προφορικού ερωτήματος. Όποιος είναι υπέρ να σηκώσει το χέρι. Ε, Κατά. Πολύ ωραία. Α, απόχεια, συγγνώμη. Κανείς δεν απέχει, επομένω ομόφωνα περνάει. Θα υποβάλουμε αυτό το ερώτημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, πάμε στο σημείο 11. Ειδικά μέτρα για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης. Η Κομισιόν προτείνει κάποιες αλλαγές στον κανονισμό 247 του 2006 για κάποια συγκεκριμένα μέτρα για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Οι βασικές αλλαγές που προτείνονται αφορούν την εισαγωγή, την επέκταση και την προσαρμογή των παρεκκλήσεων που συμφωνήθηκαν για τον τομέα της ζάχαρης και των γαλακτοκομικών προϊόντων. Ε, η διαδικασία θα αλλάξει από διαβούλευση, θα γίνει συναπόφαση μετά από την θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας την 1η Δεκεμβρίου του 2009. Ο εισηγητής είναι ο κύριος Άλβες, του δίνω το λόγο, για να μας παρουσιάσει το θέμα αυτό. Παρακαλώ. Λουίς Παόλου, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή αφορά μια τροποποίηση ισχύοντο κανονισμού που θεσπίζει παρεκκλήσεις στις ε, εξόχως απόκεντρες περιοχές από το νέο νομοθετικό πλαίσιο της ΚΟΑ. Οι εξαιρέσεις αυτές θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Πρώτου 2010. Η επιθυμία όλων των ενδιαφερομένων μερών ήταν από την αρχή να προχωρήσει η διαδικασία γρήγορα, ώστε ο κανονισμός να εγκριθεί πριν τα τέλη του έτους και να τεθεί σε ισχύ στην προβλεπόμενη ημερομηνία. Με το σκεπτικό αυτό και εγώ προσπάθησα να εκπονήσω και να δρομολογήσω την έκθεσή μου. Βέβαια, πολλά θέματα εκφεύγουν του δικού μας ελέγχου και της επιθυμία μας, γι' αυτό και η γραμματεία μας μόνο στις 2 Οκτωβρίου έλαβε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στις 26 Οκτωβρίου το έκτακτο Συμβούλιο Γεωργίας τροποποίησε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την τελευταία εβδομάδα ενημερωθήκαμε ότι το Συμβούλιο σκόπευε να επανεξετάσει αυτό το θέμα ύστερα από αίτημα της Πορτογαλίας γιατί η Πορτογαλία εξέφρασε κάποιες αφιβολίες ότι αφορά το, το νομότυπο της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το θέμα αυτό αναφέρθηκε και στο χθεσινό έκτακτο Συμβούλιο Γεωργίας όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι Όπω είπατε και εσεί, η διαδικασία αυτή θα περάσει από διαβούλευση στη συναπόφαση. Περιμένουμε λοιπόν τη νέα πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ξεκινήσουμε και τη δική μα ε, διαβούλευση. Και η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, πρόκειται να συντάξει γνωμοδότηση για το θέμα αυτό. Γι' αυτό και η Επιτροπή Γεωργίας ε, πρέπει να περιμένει τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης για να ψηφίσει τη δική τη έκθεση. Εξαιτία όλων αυτών των καθυστερήσεων θα είναι αδύνατο για μας να σεβαστούμε το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Μια και η διαδικασία θα αλλάξει και θα γίνει συναπόφαση, εξαρτώμαστε για την εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος στη νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την νομική βάση. Ε, ευχαριστώ, Λουίς Πάουλο. Ο κύριος Μάτο. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και τον εισηγητή, τον κύριο Άλβες, αλλά και τον συντονιστή ΔΕΣ, που ζήτησε εφαρμογή της απλουστευμένης διαδικασίας για την έκθεση αυτή. Κάτι που ήταν σημαντικό για να τεθεί σε εφαρμογή εμπρόθεσμα το σχέδιο. Άλλωστε θα πρέπει να περιμένουμε την 1η Δεκεμβρίου για να ισχύσει η συναπόφαση. Φυσικά θέλουμε μία νομική ασφάλεια. Θα πρέπει όλοι οι χρήστες αυτού του κανονισμού να είναι βέβαιοι για τον τρόπο εφαρμογής αυτού του κανονισμού από την 1η Πρώτου 2010, γιατί ακόμη υπάρχουν πολλές ασάφειες. Ο κύριος Άλβες μας είπε ότι την περασμένη εβδομάδα προτάθηκε επανεξέταση ορισμένων πτυχών λόγω νομικών αμφιβολιών που παρουσιάστηκαν. Εγώ δεν το είχα καταλάβει έτσι. Σε ό,τι αφορά το άρθρο 6 του κανονισμού, που είναι πολύ σημαντικό, στις 31 του μηνός, όπως ξέρετε, εξέπνει η προθεσμία του άρθρου 6, σε ό,τι αφορά τα παρασκευάσματα με βάση το γάλα που προορίζονταν για βιομηχανική μεταπίεση. Τώρα προβλέφθηκε κάποια μεταβατική περίοδος γιατί το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη με φυτικό λίπος μέχρι Τη 31 Δεκεμβρίου του 2013. Φυσικά αντιλαμβανόμαστε το σκεπτικό αυτής της διαδικασία. είναι μεταβατική αυτή η εφαρμογή και άρα δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Πάντως, θα ήθελα να σας πω ότι φυσικά υπό την επιφύλαξη των συμφερόντων του κτηνοτροφικού κλάδου, θα υποβάλω μία τροπολογία προκειμένου να καταργηθεί το χρονικό όριο της εξαίρεσης του άρθρου 6. Πιστεύουμε ότι η διάταξη αυτή δεν θα πρέπει να ισχύσει μέχρι το 2013, αλλά θα πρέπει να ισχύει επαόριστον, χωρίς χρονικό περιορισμό. Αυτά και περιμένουμε και τη συνέχιση της συζήτησης και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ελπίζω να συμφωνήσουμε όλοι και με απλουστευμένο και ταχύ τρόπο να δώσουμε μία απόφαση για να τεθεί σε ισχύ αυτό το ειδικό καθεστώς για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές που περιμένουν πώς και πώς αυτή την αναθεώρηση του κανονισμού. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μάτο. Η κυρία Πατράου Νέβες. Όντως είναι πολύ σημαντικό αυτό το έγγραφο και η τροποποίηση του κανονισμού για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Εγώ κατάγομαι από τις Αζόρες όπως και ο Λουίς Πάολο Άλβες και γι' αυτό είμαι υπέρ της εφαρμογής της απλουστευμένης διαδικασίας για τον κανονισμό αυτό. Υπήρξαν όμως κάποιες δυσκολίες για την εφαρμογή της διαδικασίας αυτής. Πάντως πρόκειται για μια έκθεση που είναι αρκετά τεχνική. Γι' αυτό και η δυνατότητα υποβολής τροπολογιών ή προστικών είναι σχετικά περιορισμένες για να μην πω σχεδόν ανύπαρκτες. Υπήρξε όμως ένα λάθος ε, ε, που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ε, κατάρτιση του εγγράφου. Θα πρέπει να γίνει ένας νέος υπολογισμός για να διορθωθεί αυτό το σφάλμα. Και να προχωρήσουμε φυσικά στη διαδικασία συναπόφασης. Σε ό,τι αφορά τη συναπόφαση, θα ήθελα να επισημάνω δύο τινά. Καταρχήν, οι ζημίες, όχι της αναβολής, γιατί θα περάσουμε από τη διαβούλευση στη συναπόφαση. Οπότε δεν μπορούμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα της 1ης του 2010, πολύ πιθανό να αναβληθεί για ένα εξάμεινο η εφαρμογή. Πάντως οι ζημίες από την καθυστέρηση αυτή δεν θα είναι σημαντικές, θα είναι περισσότερο συμβολικές. Η ενδιαφερόμενη παραγωγή για την τροποποίηση του κανονισμού θα δούμε στην αναβολή αυτή, στη μικρή παράταση, μέχρι την εφαρμογή της τροποποίησης, ε, ότι τουλάχιστον δεν λύθη άρον-άρον αυτή η απόφαση. Πάντως εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να εμπλουτίσουμε την έκθεση και να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία προκειμένου να προσθέσουμε κάποια στοιχεία που θα ευνοήσουν ακόμη περισσότερο τις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Άλλωστε η έκθεση αυτή θα είναι ένα από τα πρώτα έγγραφα που θα ε, ενταχθούν στη νέα διαδικασία της συναπόφασης. Και από αυτή την άποψη έχουμε συμφέρον να είναι εμπεριστατωμένο και καλό το έγγραφο. Και καλό έγγραφο σημαίνει λήψη υπόψη των συμφερόντων των εξόχων απόκεντρο, των εξόχως απόκεντρων περιοχών και να μην υποκύψουμε στην ανάγκη της ε, σπουδής. Αυτά και φυσικά θα έχω στενή συνεργασία ιδιαίτερα με τους συναδέλφους ε, από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Θαυμάσια. Το λόγο έχει τώρα ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελε να μας πει κάτι. Ή η κυρία Κιάρα Ιμπέριο ή ο κύριος Ατιβάμ. Ο κύριος Εριβάν. Ευχαριστώ, θα είμαι λακωνικός, γιατί βλέπω ότι πλησιάζουμε προς το τέλος της συνεδρίασής σας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φυσικά